Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα παρακαλούσα να αρχίσουμε αμέσω, αν θέλετε, με τα συμπεράσματα των ε, εισηγητών. Ποιο ε, εισηγητή ε, θέλει να αρχίσει, Ποιο έχει σειρά πρώτο, Ευχαριστώ πολύ τους αγαπητούς συναδέλφους των μέσων ενημέρωσης. Μερσή μποκού και χαίρετε. Καλή σας μέρα. Αλλά εσύ πρώτος, η Σάρον Μπόλς, δεν ξέρω, αποφασίστε. Κύριε Μπόλς, παρακαλώ. Σα ε, Σας ευχαριστώ. <clears throat> Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε δύο τμήματα στη συνεδρίαση. Καταρχήν, ποιος θα χαράξει το δρόμο για την ανάκαμψη και το δεύτερο κομμάτι για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να οχυρώσουμε μέσα στην Ευρώπη το δρόμο για την ανάκαμψη. Ο στόχος μας ήταν να δούμε ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρείται αυτή τη στιγμή από πολλού ότι υπάρχει μια έλλειψη δημοκρατική νομιμοποίηση όταν λαμβάνονται όλε οι αποφάσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στο επίπεδο των εθνικών κρατών και αυτό οδηγεί σε μεγάλη απογοήτευση για πολλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σε θεώρησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να ψάξουν να βρουν τρόπου για να βελτιώσουν τη συμμετοχή του στι διαδικασίε αυτέ, ώστε <clears throat> μεταξύ άλλων να εξασφαλίσουν και μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα, νομιμοποίηση και αποτελεσματικότητα και να σέβονται το ρόλο ημέν των δε. Και αυτό υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα από τους κοινοβουλευτικούς από τα έξι ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα τελικά συμπεράσματα αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί η δημοκρατική λογοδοσία μέσα σε μια διαδικασία συνεργασίας μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Η συζήτηση βέβαια θα συνεχιστεί στην συνεδρίαση που θα οργανώσει η Κυπριακή Βουλή τον Απρίλιο στη Λευκοσία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι μπορούμε μέσα στη συζήτηση αυτή να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των δημοσίων αγαθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μπορέσουν να καλύπτονται από ένα ποσοστό του προϋπολογισμού 2 με 3% και θα πρέπει να συζητηθεί και το ποιος θα επομίζεται τις ζημίες και ποιος θα καρπούται τα ωφέλη. Πρέπει λοιπόν τα θέματα των ευρωπαϊκών κοινών αγαθών να αντιμετωπιστούν στη δεύτερη πλευρά της ε, συζήτησης που ήταν η αντιπαράθεση της ανάπτυξης με τη λιτότητα. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με δύο ομιλητές έξω από το Κοινοβούλιο που παρουσίασαν ενδιαφέρουσες απόψεις. Είχαν ίσως σαν στόχο να είναι προκλητικοί και όχι απλώς να δημιουργήσουν μια συνένεση στον χαμηλότερο κοινό παρανομαστή. Συμφώνησαν ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία συνεχίζεται η κρίση. Ο κύριος Σιμ θεώρησε ότι μόνο από τη λιτότητα μπορεί να προκύψει η ανάκαμψη, ενώ πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες είπε υποστηρίζουν την ανάκαμψη. Οι χώρες οι οποίες έχουν ε, μεγάλα προβλήματα είναι οι χώρες οι οποίες χρηματοδότησαν την ανάπτυξή τους στο παρελθόν με υπερχρέωση. Αυτό δεν είναι η λύση γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εσωτερικής ανταγωνιστικότητας και όχι μονάχα μια προσωρινή έλλειψη ζήτηση. Ο κύριος Τίμπερ, ο δεύτερος ομιλητής είπε ότι με την κρίση αυτή και επειδή είναι μάλλον ζωφερό το οικονομικό σκηνικό, η λιτότητα προκάλεσε μεγαλύτερη ύφεση και δεν τη θεράπευσε την ύφεση. Αντίθετα θεωρεί ότι θα ήταν ε, σημαντικό να μην είμαστε υπερβολικοί στην μείωση των ελλημάτων. Υπήρξαν λοιπόν διαφορετικές προτάσεις σε σχέση με την έννοια της χώρας προέλευσης. Αλλά οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων μαζί με τους κοινοβουλευτικούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησαν τις διάφορες επιλογές σε σχέση με την κατάσταση της χώρας τους και τόνισαν την ανάγκη να γίνει πιο αντιληπτή η ανάγκη για δημοκρατική λογοθεσία στα πλαίσια των θεμα... θεμάτων αυτών. Και έτσι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητηθούν πολύ σημαντικά θέματα τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο και τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως η ανάπτυξη και το δημόσιο χρέος. <coughs> Ευχαριστώ πολύ. Όλα, ολά μας Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συζητήσαμε για δύο ώρες όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και των Εθνικών Προϋπολογισμών. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι η συνεδρίαση αυτή ήταν επιτυχής ε, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Είχαν εγγραφεί 103 μέλη εθνικών κοινοβουλίων. Αντιπροσωπεύονταν όλα τα κράτη-μέλη εκτός από τη Σλοβακία για κάποιο λόγο εθνικής σημασίας. Τέσσερις πρόεδροι εθνικών κοινοβουλίων και αρκετοί πρόεδροι επιτροπών. Τι προτείναμε στα εθνικά κοινοβούλια να προσπαθούμε κάθε χρόνο να βρίσκουμε μια εβδομάδα ή μισή εβδομάδα κατά την οποία θα συναντώμαστε όλοι. Αυτή θα ήταν η επιθυμία μας. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε να προσδίδουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση στην εθνική συζήτηση περί προϋπολογισμού. Θα επιτρέπει την ένταξη του εθνικού διαλόγου, της εθνικής συζήτησης ε, στον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό, ώστε να είμαστε επικοδομητικοί για το μέλλον. Τον οποίο χαιρετίζω είχε πει κάποια στιγμή λυπημένος δεν έχω το αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχω κάποιον συνομιλητή διακοινοβουλευτικό και ουσιαστικά ο διακοινοβουλευτικός ε, συνομιλητής είναι ουσιαστικά η συνέλευση που εμείς εκπροσωπούμε σήμερα το πρωί όσον αφορά το περιεχόμενο του κοινοτικού προϋπολογισμού οι εθνικές προσδοκίες από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ακούσαμε διάφορες απόψεις ανάλογα με τη χώρα για διάφορα θέματα όπως η γεωργία, τα διαρθρωτικά ταμεία. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον ήταν ότι διαπιστώνουμε τις προσπάθειες εμβάθυνσης ε, της έννοιας της προστιθέμενης αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν δίνουμε περισσότερα χρήματα ή αφαιρούμε περισσότερα χρήματα από μια χώρα Αυτά δεν είναι απλά περισσότερα χρήματα, είναι περισσότερα ευρωπαϊκά χρήματα που προέρχονται από τους φορολογούμενους των άλλων χωρών. Τι κάνουμε με αυτά τα χρήματα και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τον προϋπολογισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλοί επέμειναν και αυτό θα ευχαριστήσει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε τα μέσα εκπαίδευσης, κατάρτισης, επένδυσης, μακροπρόθεσμης. Ο πρόεδρος Μπαρόσο επιμένει πάντα αυτά είναι θέματα που δεν έχουν ψηφοφόρους. Όπως είπαν και οι αντιπρόσωποι της Ιρλανδικής Προεδρίας ε, στις χώρες όπου είναι σημαντικό κατά τα μία συνοχής ε, αυτό θα βοηθήσει να επιστρέψει στην ανταγωνιστικότητα και αυτό βασίζεται και σε, αυτούς τους, ε, σε αυτά τα κονδύλια. Η Ιρλανδία για παράδειγμα καταφέρνει να ε, αφιερώσει 40% των ταμείων έρευνας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά οι χώρες της πολιτικής συνοχής και ειδικά οι χώρες υπό πρόγραμμα αρρωγής είπαν ότι τα εθνικά ε, προγράμματα προσαρμογής ε, εξαντλούν ε, τα προγράμματα ανάπτυξης. Δέκα χώρες για τις οποίες τα ταμεία συνοχής αποτελούν το 1 τρίτο των δημόσιων επενδύσεων και άλλες χώρες τις οποίες δεν προσωπεύουν τα 2 τρίτα. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτές τις χώρες ακριβώς τη στιγμή όπου κάνουν τόσο μεγάλες προσπάθειες. Τέλος, με ενδιαφέρον ακούσαμε έναν εκπρόσωπο ενός σημαντικού πολιτικού κομμάτου μιας μεγάλης ε, ευρωπαϊκής χώρας, ε, χώρας που πάντα προσέχει τη δημοσιονομική αυστηρότητα είπε ότι ένας καλός προϋπολογισμός της Ευρώπης μπορεί να βοηθήσει εξυγίανση των εθνικών προϋπολογισμών, τη μείωση ορισμένων ε, δαπανών χάρη στην αμοιβαιοποίηση. Έχουμε την, την εξωτερική πολιτική ε, μέσω της κυρίας Άστον. Εκεί μπορούμε να μειώσουμε κάποια εθνικά δίκτυα. Το ίδιο ισχύει και σε θέματα τελωνίων, σε θέματα ε, σύνοριοφυλάκων. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα για την επόμενη χρονιά. Να δούμε τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες, χαμηλότερες δαπάνες με περισσότερα αμοιβαιοποίηση. Δύο τελευταία λόγια για τους πόρους. Θα θέλαμε επίσης, θέλαμε να μάθουμε πώς έβλεπαν τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού οι εθνικοί βουλευτές και πώς θα χρεώνονται οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Γι' αυτό λίγα ακούσαμε. Ακούσαμε από φίλους του Ολλανδικού Κοινοβουλίου να μας υπενθυμίζουν ότι η υλοποίηση του φόρου περί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα μπορούσε να ελαφρύνει τη συμβολή αυτών των χωρών εφόσον δεχθούν την αρχή αντιστοιχέ ενό κομματιού αυτών των πόρων στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Επ' αυτού ανακοινώνω ότι στη συζήτηση του 2014 για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό που θα οργανίσουμε τον επόμενο Οκτώβριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, η Επιτροπή Προπολογισμού για πρώτη φορά θα προτείνει η συζήτηση να αφορά όχι μόνο τις δαπάνες αλλά και τα έσοδα και θα πούμε χώρα προς χώρα ποιος πληρώνει τι για τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού, ποια είναι τα προβλήματα, ποιοι είναι οι προνομιούχοι του τρέχοντος συστήματος και ποιοι είναι εντό αγωγικών θύματα του σημερινού συστήματος χρηματοδότησης. Έτσι ελπίζουμε να προχωρήσει η συζήτηση να παρέχουμε επιχειρηματολογία ενώπιον των Εθνικών Κοινοβουλίων για την επεξεργασία των δικών τους προπολογισμού, ώστε να δουν μαζί μας τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Ευχαριστώ, αλλά υπερβάσπερες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε του Κοινοβουλίου, ε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνάντηση, για αυτό το ραντεβού μας θα έλεγα, γιατί μετά τη θέση σε ισχύ του Δημοσιονομικού Συμφώνου, η φετινή εμπειρία αποδείχθηκε πολύ διαφορετική από εκείνη ε, των παρελθόν ετών για δύο λόγους. Πρώτον, ο Λέλα Μασούρα ανέφερε μόλις συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Αλλά αισθανθήκαμε ένα είδος και επίπεδο συμμετοχής πολύ διαφορετικό από εκείνα που είχαμε φανταστεί ως σχήματα πριν τη θέση σε του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Και αυτό το λέγω και ε, σε ό,τι αφορά τους ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν λάμπουν για τις παρουσίες τους καθώς ε, είναι στην έδρα τους ε, η συνεδρίαση. Φέτος ε, ήταν πολύ μεγάλη προσέλευση των Ευρωβουλευτών και τα παράλληλα εργαστήρια είναι μια φόρμουλα που δεν μας επέτρεψε βέβαια να καταλήξουμε σε κοινέ θέσει, γιατί δεν είναι αυτός ο προορισμός μας να πονήσουμε κοινά κείμενα αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένες οι ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών και εντός των διαφόρων πολιτικών οικογενειών είχαμε την ίδια αίσθηση τη Δευτέρα το απόγευμα. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ε, χωρίσαμε τις εργασίες, μοιράσαμε σε δύο ε, συνεδριάσεις. Η πρώτη αφορούσε ε, την ανεργία των νέων με ένα πάνελ πέντε εμπειρογνωμόνων βουλευτών, όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω. Ο συνάδελφος Ασπύρος από την Ισπανία συνάδελφος Κρεμαστινός από την Ελλάδα και η κυρία Φίλατοφ ε, της Φιλανδίας ε, παρουσίασαν την κατάσταση ως προς την ε, απασχόληση των νέων στη χώρα τους και η κυρία Φίλατοφ μας περιέγραψε πάρα πολύ συγκεκριμένα το μηχανισμό για την εγγύηση προς τους νέους, εγγύηση για την νεολαία που ισχύει στη Φιλανδία. Αυτή η στρογγυλή τράπεζα, σε αντίθεση με την επόμενη, συγκέντρωσε βουλευτές από κάθε γωνιά της Ευρώπης, Βόρεια, Νότο, Ανατολή, Δύση, χωρίς καμία ε, διχογνωμία ή απόσταση απόψεων. Η πρώτη διαπίστωση λοιπόν είναι ότι υπάρχει ευρεία πολιτική συνένεση για να πούμε ότι με τον ίδιο τρόπο που θέλουμε να καταπολεμήσουμε την καταστροφή και τη σπατάλη στο περιβάλλον, θα πρέπει ε, να ε, καταπολεμήσουμε και αυτού του είδου τη σπατάλη στο ανθρώπινο δυναμικό, να μην αφήσουμε να πάει χαμένη μια γενιά χωρίς πρόσβαση στην αγορά εργασία. Υπάρχουν εμπειρίε λοιπόν που ε, στη Φιλανδία, στην Αυστρία, στο Λουξεμβούργο αλλά και στη Γαλλία σήμερα έχουν υιοθετηθεί και το είπαν και οι Γερμανοί συνάδελφοι. Αντίστοιχα επίση με το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, παράλληλα με την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχαμε και πρωτοβουλίε στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αντίστοιχα λοιπόν ε, για την αγγίηση, για την νεολαία, θα μπορούσαμε έτσι να συγκλίνουμε ε, και να καταλήξουμε σε μια πολιτική ευθύνη στα Κοινοβούλια. Το δεύτερο είναι το θέμα το πάγιο, πώς συνδέεται η οικονομία με τα κοινωνικά. Το άρθρο 9 της Συνθήκης Λισαβόνας ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ, διότι ε, ανάγεται ε, σε ένα υπόλοιπο, αν θέλετε, της οικονομίας ε, η κοινωνική διάσταση, ενώ θα πρέπει να είναι προτεραιότητα τα κοινωνικά θέματα και να καθορίζουν και τις υπόλοιπες πολιτικές. Τρίτον, έγινε μια συζήτηση για να δούμε κατά πόσο η ενεργεία των νέων αφορά τους νέους χωρίς προσόντα τους, ανειδίκευτους ή όχι καταλήξαμε ότι υπάρχουν μεν οι αντιδικευτοί που είναι σκέτη φρίκη, αλλά δεν θα πρέπει αυτό το δέντρο να, να κρύψει το άλλο δέντρο του δάσους που είναι οι νέοι με δεξιότητε και προσόντα που στις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες δεν βρίσκουν παρόλα αυτά δουλειά. Επόμενη παρατήρηση. Θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε την ετήσια έκθεση για την ε, ε, απασχόληση για να φροντίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαγρυπνεί ε, ταυτόχρονα με την κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης να καταθέτουν τα κράτη-μέλη και ένα σχέδιο για την απασχόληση και για την εγγύηση για τους νέους. Μια τελευταία παρατήρηση που έκανε μια Σουηδή συνάδελφος να υποχρεωθούμε να δεσμευτεί το Συμβούλιο να μην μειώσει τις εγγύησεις για την νεολαία ε, ούτε ως προς την πρικοδότηση ούτε ως προς τη διάρκεια γιατί ορισμένοι θεωρούν ότι αντί για ένα τετράμινο θα χρειαστεί εξάμινο για αυτή την υπόθεση. Το είπε πολύ ωραία η συνάδελφος από τη Σουηδία και με βάση την φιλανδική εμπειρία. Ε, όταν είσαι νέος το τετράμινο έχει σημασία γιατί ε, αυτό κάνει τη διαφορά. Ε, για το κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν τα προγράμματα προσαρμογής των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσκολίες, είχαμε και εκεί ε, ειδικού εκπροσώπους εμπειρογνώμονες και ακολούθησε συζήτηση και αυτό ήταν χαρακτηριστικό ε, που μίλησαν κυρίως οι χώρες που και οι συνάδελφοι είναι από χώρες σε μνημόνια. Ο συνάδελφος ε, από την ε, από τη Λετωνία ε, μας μίλησε για την πολιτική συνοχή που ανέφερε προηγουμένως και ο ε, Λαμασού και πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν τα προγράμματα και επενδύσεις. Και στη συνέχεια τα αποτελέσματα της Λετωνία τα γνωρίζουν όλοι, αλλά ε, το τόνισε και ο ίδιο, σήμαινε μια μετανάστευση 10% ε, του πληθυσμού και κυρίως των νέων. Τα συμπεράσματα της Στρογγυλής Τράπεζας ήταν κυρίως η ανάγκη στα προγράμματα προσαρμογής να συμμετέχουν οι εταίροι, είτε αυτή είναι η κοινωνική εταίροι, είτε τα εθνικά κοινοβούλια. Υπάρχει μια δυσκολία, όσο και μια αντίφαση ε, στα προγράμματα και τα μνημόνια, διότι ξυλώνουν τον, τους αυτόματους σταθεροποιητές που είναι από τα ατού της ευρωπαϊκής οικονομίας ή ήταν στην αρχή της κρίσης. Από πλευράς μου τόνισα την πάγια θέση του Κοινοβουλίου ή ε, τουλάχιστον της Επιτροπής μου. Θεωρούμε ότι η Τρόικα θα πρέπει να γίνει τετραμερής να συμμετέχει και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ε, στα προγράμματα και τα μνημόνια. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι όλη η συζήτηση που γίνεται για τους λεγόμενους πολλαπλασιαστές των πολιτικών ε, λιτότητας. Είπαμε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο αυτό το ζήτημα ε, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές πολιτικές που υιοθετούνται και θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου θα πρέπει να είναι ένα συμβούλιο που θα πρέπει να ασχοληθεί με τον αντίκτυπο των πολιτικών λιτότητας. Να είναι ευρωπαϊκή απάντηση για όλη την Ευρώπη και όχι ε, προϊόν ε, διμερούς ε, διαπραγμάτευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων. Μιλήσαμε για την ετήσια εξέταση της ανάπτυξης θα πρέπει να το συζητήσουμε και στα πλαίσια ε, ε, του πολιετούς ε, προγράμματος, δημοσιονομικού πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από το 25% που είναι για μας ιερό. Ευχαριστώ κυρία Μπερές, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο. Ο ο κύριος Παρόσο ε, θα κάνει την ε, ομιλία του, αλλά μετά πρέπει να φύγει γιατί στις 10 η ώρα αρχίζει η συνεδρίαση της Κομισιόν. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Φανρομπάη και με τον πρόεδρο του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Σας παρακαλώ λοιπόν να είσαστε σύντομοι στο μέλλον. Ο κύριος Μπαρόσο. Πρόεδρε Σούλτς, πρόεδρε Φανρομπάη, <coughs> πρόεδρε της ε, Βουλής Ιρλανδίας. Κυρίες και κύριοι, <clears throat> εισήγητέ, κυρία Μπάουλ, ε, μπερέ, κυρία Λαμασούρ, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ όλους και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα έχει γίνει ένα αναπόσπαστο στοιχείο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε στο διακοινοβουλευτικό διάλογο και στο μέλλον. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να φύγω σύντομα γιατί ήδη έχω καθυστερήσει την ε, συνεδρίαση της Κομισιόν μέχρι τις 10 για να μπορέσω να συμμετάσχω στην ενακτήριά σας συνεδρίαση. Αλλά ο κύριος Μάρος Σεύκοβιτς, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος για τα διαθεσμικά θέματα με τα με το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα είναι παρόν σε όλη τη διάρκεια τη συνάντησή σα Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρισκόμαστε στο Σταυροδρόμι σήμερα και προχωρούμε προ την εμβάθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε αυτό αν θέλουμε η Ευρώπη να βγει από την κρίση και να προχωρήσει προ ένα πιο σταθερό και βιώσιμο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να κινούμεθα προς την κατεύθυνση ενός πραγματικού ευρωπαϊκού δημοσίου χώρου. Ναι, πρέπει να γίνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να το κάνουμε αυτό με την υποστήριξη των πολιτών μας, με δημοκρατική ε, συζήτηση και με δημοκρατική νομιμοποίηση. Για μένα η δημοκρατία είναι κάτι το απαράγραπτο και το εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Από την αρχή της κρίσης και έχουμε αντιμετωπίσει πολλές από τις αδυναμίες της Ευρώπης, έχουμε ενισχύσει τις οικονομίες της Ευρώπης, έχουμε βοηθήσει την οικονομική διακυβέρνηση και έχουμε αντιμετωπίσει πολλές από τις προκλήσεις ενώπιών μας. Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι αυτοί οι οποίοι περίμεναν να καταρρεύσει το ευρώ αποδείχθηκαν ότι είχαν λάθος. Έχει εξασφαλιστεί η επιβίωση του ευρώ και από το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ζώνη του ευρώ ε, από το 2012 συγγνώμη, αρχίζουμε να βγαίνουμε από την ύφεση. Οι οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται και αυτό οφείλεται και στι εξελίξεις που αφορούν τη μελλοντική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μονάχα στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων. Επομένως, το πρώτο πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι οι προσπάθειες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο δεν είναι μάταιες, είναι ιδιαίτερα λυσιτελείς αντίθετα. Αυτό είναι το επόμενο μήνυμά μου. Και πάλι με την ίδια έμφαση θέλω να το τονίσω, δεν υπάρχει καθόλου περιθώριο για να επαναπευόμαστε. Η κοινωνική κατάσταση είναι ιδιαίτερα οξία στην Ευρώπη. Η ανεργία, ιδίω η ανεργία των νέων, είναι μια τεράστια ανησυχία για όλου μα. <clears throat> Σε 12 από τα 27 κράτη-μέλη μα η ανεργία των νέων ξεπερνάει το 25% σε κάποια κράτη-μέλη μας, όπως ε, έχω τονίσει και πολύ σαφώς, αντιμετωπίζουν ένα πραγματικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης σε κοινωνικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια έχουν κατανοήσει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρουμε ότι πολλά από τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της ανεργίας βρίσκονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά δεν μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Ήδη το 2009 είχα αναλάβει μια πρωτοβουλία για μια διάσκεψη κορυφή για την απασχόληση σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Δεν ήταν πολύ θετική τότε η απόκριση, για να είμαι ειλικρινή. Ήταν μια απογοήτευση. Μόνο μερικά κρατημέλη δέχτηκαν να παρασταθούν σε αυτή τη διάσκεψη κορυφής και αυτή η διάσκεψη έγινε κατά κάποιο τρόπο μια διάσκεψη κορυφής μεταξύ δύο κρατών μελών μονάχα. Δεν μπορούμε όμως να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω. Να έχουμε ομάδες δράσης για να αντιμετωπίσουμε τα 8 κράτη-μέλη που είναι ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και να κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έχουμε προτείνει την ε, λεγόμενη εγγύηση για τους νέους. Ελπίζω ότι θα εγκριθεί αυτή η ρύθμιση Χρειάζεται όμως να έχουμε και περισσότερα μέτρα κατά της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων. Έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανεργίας των νέων εγκαίρως μέσα στα πλαίσια της συζήτησης για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν υπάρξει πολιτική θέληση και τα κατάλληλα εργαλεία μπορούμε να το πράξουμε αυτό η πρώτη μας προτεραιότητα στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να είναι οι πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο της επόμενης εβδομάδας. Οι προοπτικές αυτές είναι ένα απαράγραπτο τμήμα της απάντησής μας στην οικονομική κρίση. Είναι απαραίτητε αυτέ οι προοπτικέ για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τι επενδύσει και ιδίω στι πιο ευάλωτε περιοχέ και χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρά το γεγονό ότι υπάρχει η πτυχή τη αλληλεγγύη στι πολιετή αυτέ προοπτικέ, δεν είναι μονάχα χρήματα για του φτωχότερου, για τι λεγότερο ευμαρεί περιοχέ. Όλε οι χώρε είναι καθαροί αποδέκτε από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, όπως νομίζω ότι έγινε σαφές και κατά τη διάρκεια των συζητήσεών σας. Ακόμα και οι μεγαλύτερες και πιο δυνατές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν μια υποστήριξη για τις υποδομές, για τις επενδύσεις τους από τις δημοσιονομικές προοπτικές και αντλούν ωφέλη από αυτά τα χρήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κυβερνήσει οι οποίε μιλάνε για την υποστήριξη τη ανάπτυξη και τη ανταγωνιστικότητα, σωστά και στι δύο περιπτώσει, αλλά μετά όταν έρχονται στι συζητήσει του πιο σημαντικού εργαλείου που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσουμε τι επενδύσει, κάπου βάζουν νερό στο κρασί του. Εγώ δεν έχω χάσει κάθε ελπίδα για τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές παρά την πίεση που ασκήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει και αυτό ένα σημαντικό ρόλο για την επίτευξη μιας σωστής συμβαστικής λύσης. Επίσης θα πρέπει να περατώσουμε την νομοθεσία για την ενιαία εποπτική αρχή για τις τράπεζες. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε περισσότερο σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Ε, η δημιουργία του μηχανισμού του ESM, του συστήματος ε, σταθερότητας για το τραπεζικό σύστημα. Χρειαζόμαστε όμως και ένα τώρα ενιαίο μηχανισμό επίλυσης για τα τραπεζικά ιδρύματα και η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια πρόταση για τα θέματα αυτά πριν από το καλοκαίρι. Πρέπει επίσης να περατωθεί η διαδικασία για το λεγόμενο TUPAC, το δίπτυχο που είναι η απαραίτητη νομοθεσία για την οικονομική διακυβέρνηση. Είναι και μια δοκιμασία αξιοπιστίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, θέλω να σα ευχαριστήσω για αυτή την εκδήλωση και ιδίω στα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που ήρθαν στι Βρυξέλλε για να συζητήσουν για τι πτυχέ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, <clears throat> που είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την οικονομική διακυβέρνηση και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών μα. <clears throat> Έχετε συζητήσει λοιπόν τι προτεραιότητε αυτέ <clears throat> που έχει θεσπίσει η Κομισιόν στην ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη <clears throat> για το 2013. Πρέπει να ξεπεράσουμε και αυτό το θέμα. Εάν θέλουμε να επιστρέψουμε σε πραγματική ανάπτυξη, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε τρία κύρια μέτωπα. Πρώτα, μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη. Με το να γίνουν οι απαραίτητε διαρθρωτικέ αλλαγέ που θα επιτρέψουν να ξαναβρούν την οικονομική ισορροπία του και να αυξήσουν την αναγωνιστικότητα των οικονομιών του. <clears throat> Εδώ κοινή μας εστίαση θα πρέπει να είναι οι μεταρρυθμίσεις για πιο ευέλικτη αγορά εργασίας και πιο ευέλικτες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι κεφαλαιόδη για την ανταγωνιστικότητα. Και επίσης πρέπει να δώσουμε έμφαση σε όλους τους τομείς υποδομών, ενέργεια, ψηφιακή οικονομία, μεταφορές και αυτά περιλαμβάνονται στην ετήσια ε, επισκόπηση για την ανάπτυξη. Επίσης θα πρέπει να πάρουμε τις απαραίτητες δράσεις για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών προϋπολογισμού των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν τα 27, σύντομα 28 κράτη-μέλη με το να αυξήσουν την λογοδοσία και τους μηχανισμούς επίσης αλληλεγγύης θα μπορέσουν να ενισχύσουν την οικονομική ένωση και να συνεχίσουν και την πορεία προς μια πολιτική ένωση με μεγαλύτερο διασταυρούμενο έλεγχο και δημοκρατικό έλεγχο όλων των ε, αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση της Κομισιόν για την γνήσια οικονομική και πολιτική ένωση που παρουσιάστηκαν από την Κομισιόν αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ και θέτει το ερώτημα του πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και να την οδηγήσουμε σε μεγαλύτερη ενσωμάτωση και ολοκλήρωση στον χρηματοπιστωτικό, οικονομικό αλλά και πολιτικό χώρο. Δίνει κάποιες προτάσεις και κάποιες εμπνεύσει, κάποιε από τι οποίε είναι πιο βραχυπρόθεσμε, κάποιε πιο μακρόπνοε. Κάποιε από αυτέ εξαρτώνται μόνο από την πολιτική θέληση, μπορούν να γίνουν και τώρα. Άλλε απαιτούν αλλαγή των συνδικών. Σε όλε τι περιπτώσει όμω χρειάζεται μια σε βάθο προβληματική και ανταλλαγή απόψεων σε πολιτικό επίπεδο. Η κρίση των τελευταίων ετών κατέδειξε ποια είναι τα όρια των μεμονωμένων δράσεων σε επίπεδο κράτου μέλου. Και επίση την ανάγκη για ευρωπαϊκή συνεργασία και ολοκλήρωση πολλές φορές οι λύσεις που προκρίθηκαν ήταν λύσεις ad hoc. Τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν μια έκτακτη κατάσταση, χρειάστηκε να έχουν πυροσβεστικές προσπάθειες και συγχρόνως ενώ έσβηναν τη φωτιά να χτίζουν. Αυτό κάνουμε ακόμα σήμερα. Αλλά θα πρέπει συγχρόνως να λάβουμε υπόψη την ανάγκη να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία, τη λογοδοσία και την ε, διαφάνεια παράλληλα με όλε τι προσπάθειε που καταβάλλονται για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και, το Εθνικό, και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει πάντα ένα σύστημα διακυβέρνηση το οποίο είναι πολυεπίπεδο. Η μέγιστη δημοκρατική λογοδοσία λοιπόν θα πρέπει να δίδεται στο επίπεδο που λαμβάνονται οι αποφάσει, λαμβάνοντα υπόψη την αλληλοσύνδεση όλων των επιπέδων όπου οι αποφάσει αυτέ θα έχουν επίπτωση. Αυτό σημαίνει, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, ότι η δημοκρατική λογοθεσία και η νομιμοποίηση στην Ευρώπη του 21ου αιώνα θα πρέπει να λαμβάνει χώρα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται ως παίγνιον μηδενικού αθροίσματος. Είναι συμπληρωματικές αυτές οι δύο πλευρές. Η κοινοβουλευτική διάσταση είναι ακριβώς ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να παίξει το ρόλο του και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και εδώ διακυβεύονται πάρα πολλά θέματα. Οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται και να προετοιμάζονται με τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και στα δημοσιονομικά θέματα και στα θέματα του προπολογισμού και στα μικρο, μακροοικονομικά ζητήματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τον οικονομικό αυτό διάλογο όπως προβλέπεται από την νομοθεσία του εξάπτυχου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη μια πλευρά της Κομισιόν, του Συμβουλίου και της Ευρωομάδας πρέπει να εμπλέξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πριν από τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης και πριν από την έγκριση των ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων. Η Κομισιό και το Συμβούλιο επίσης θα πρέπει να παρίστανται σε συναντήσεις συστηματικά των ε, εθνικών κοινοβουλίων και να λαμβάνει υπόψη και τις προτάσεις που προέρχονται και από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εν γέννη λοιπόν μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση ζητά μια κοινή προσέγγιση για το μέλλον της ένωσης αυτής. Αυτό είναι πολιτικά σαφές. Θα πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα. Είναι κατάλληλη στιγμή τώρα μια προεκλογική εκστρατεία είναι και η πιο πρόσφερη στιγμή και σκέφτομαι στις εκλογές του 2014 να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στο λαό με ευρύτερη συζήτηση και καλύτερη αντίληψη του τι διακυβεύεται. Και αυτό μπορούμε να το πράξουμε με το να ενισχύσουμε τα, τους φορείς της πολιτικής, με το να ενισχύσουμε τον ρόλο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Γι' αυτό η Κομισιόν έχει προτείνει να υπάρξει ευρωπαϊκό καθεστώς νομικού χαρακτήρα στα πολιτικά κόμματα, γιατί θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό τα ευρωπαϊκά κόμματα θα δώσουν πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα στις εκλογές, ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε σε μια δημοκρατική ευρωπαϊκή συζήτηση. Κλείνω, αγαπητά μέλη, λέγοντάς σας ότι βαθμία, βήμα-βήμα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις προκλήσεις ενωπιών της με επιτυχή τρόπο. Παραμένουν πολλές ακόμα προκλήσεις, ιδίως στον κοινωνικό τομέα, αλλά επιτυχάνουμε πρόοδο και αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα διαρθωτικού χαρακτήρα και προβλήματα εμπιστοσύνη. Αυτοί οι οποίοι είχαν μιζάρι στην αποτυχία του ευρώ έχουν χάσει το παιχνίδι. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε ότι είχαν λάθος και δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να πάψουμε τις προσπάθειές μας στο ευρώ τη στιγμή που αρχίζει η πορεία αυτή η κοινή με το ευρώ να αποδίδει καρπού. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Δεν αρκούν μονάχα τα συγκεκριμένα κίνητρα που δίδονται εδώ και εκεί θα πρέπει να δώσουμε μια σαφή εικόνα προόδου και στις αγορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω ότι πρέπει τώρα να φύγετε τρέχοντα. Το λόγο έχει τώρα ο πρόεδρο του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Φαρόμπερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής και αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση παρευρίσκομαι σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος ε, και ως πρώην πρόεδρος Εθνικού Κοινοβουλίου που έχω την ευκαιρία να σας συναντήσω στην αρχή αυτού του νέου έτους. Το 2013 ξεκίνησε πιο ελπιδοφόρο τόσο για την Ευρωζώνη όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις και το ανέφερε ήδη ο πρόεδρος της Επιτροπής ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Είναι πλέον σαφές ότι το ευρώ είναι μία, αναστρέψιμο πρόγραμμα. Οι χώρες που δέχτηκαν πιέσει ε, από τις αγορές όπως Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, εκεί τα δημοσιονομικά φαίνονται καλύτερα, αυξάνονται οι εξαγωγές και από την οικονομική πλευρά τα spreads μειώνονται και ο δημοσιονομικός κατακαιρματισμός ε, σιγά σιγά απαλήφεται. Όλα αυτά είναι ελπιδοφόρες ενδείξεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Εξάλλου βρισκόμαστε σε μια διαδικασία υπέρβασης μιας από τις μεγαλύτερες οικονομικές υφέσεις ε, τις μεγαλύτερες ουσιαστικά από τη δεκαετία του 30, όπου γνωρίσαμε μια υπαρξιακή κρίση του ευρώ. Μια κρίση που έκανε τους ανθρώπους να φοβούνται για τις αποταμιεύσεις τους και να έχουν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την επιβίωση του ίδιου του νομισματός τους. Τίποτα δεν θα μπορούσε να έχει καταστρέψει τόσο πολύ την εμπιστοσύνη στο όλο σύστημα Ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Η σταθεροποίηση της ε, Ευρωζώνης αποτέλεσε προτεραιότητα για εμάς τα τελευταία τρία χρόνια για έναν πολύ απλό λόγο. Χωρίς τη σταθερότητα αυτή δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, δεν, μπορεί, δεν μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασία. Από αυτή την άποψη, το 2012 θα θεωρείται σημείο καμπής. έγινε τεράστιος όγκος εργασίας στα κράτη-μέλη, στην Ευρωζώνη και στο σύνολο της Ένωσης. Μόνο αφού περάσουν αυτές οι δύσκολες στιγμές ε, θα αντιληφθούν οι άνθρωποι πόσο δρόμο έχουμε καλύψει. Και δύο κατευθυντήρες αρχές ε, οδήγησαν όλες τις αποφάσεις που λάβαμε μεγαλύτερη ευθύνη, λογοδοσία και μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Και αυτά τα δύο είναι αλληλοσυνδεόμενα μεγαλύτερη λογοδοσία για τι εθνικέ κυβερνήσει, όπω η σύναψη της, ε, του Δημοσιονομικού Συμφώνου που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές ε, αυτού του μήνα και την θαραλέα υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είναι σκληρέ μεν αλλά αναγκαίε και μεγαλύτερη αλληλεγγύη ειδικότερα με την καθιέρωση ενός μόνιμου ταμείου διάσωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα για την προστασία των οικονομιών μα από μεγάλης κλίμακας οικονομικές ε, και χρηματοοικονομικές κρίσεις. Προοδεύσαμε στον οικονομικό συντονισμό και στην Τραπεζική Ένωση. Αυτά τα βήματα συνέβαλαν σημαντικά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, στην αντοχή και την ακαιρεότητα της Ευρωζώνης. Προχωρήσαμε δεχόμενη πίεση και πιέσεις από τις ε, χρηματαγορές, αλλά ακόμη και χωρίς αυτές τις πιέσεις θα ήταν αναπόφευκτες αυτές οι ρυθμίσεις, ούτως ή άλλως. Είτε, με, είτε χωρίς το ευρώ, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αργά ή γρήγορα θα καθίσταν το απαραίτητες, όχι μόνο λόγω των πιέσεων από τις αγορές. Οι αγορές δεν είναι πάντα λογικές, αλλά διότι αντικειμενικά είναι παράγοντες που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε η βιωσιμότητα του χρέους, η ανταγωνιστικότητα, οι δημογραφικές αλλαγές και ούτω καθεξής. Είναι απλά αδύνατον να συσσωρεύουμε διαδοχικά διψήφια ελλείμματα στους προπολογισμού χωρών, στους τρέχοντες λογαριασμούς, στο ισοζύγιο πληρωμών, χωρίς καμία συνέπεια. Είναι σαν να θέτουμε σε κίνδυνο το μέλλον των λαών μας. Αν είχαμε αντιδράσει έγκαιρα πριν από 10 χρόνια, θα είχαμε αποφύγει πολλές από τις δυσκολίες, πολλά από τα προβλήματα. Αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολη είναι η προσαρμογή, αλλά αρχίζουν με να βλέπουμε αποτελέσματα βελτίωσης. Σήμερα η πρόκλησή μας είναι ότι με την επαναφορά της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης ουσιαστικών παραγόντων υπάρχει πάντα κάποια σύνδεση μεταξύ, υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ της επιστροφής της σταθερότητας και της ε, εκ νέου ανάπτυξης. και στη συνέχεια με την αύξηση της απασχόλησης. Πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στο να μειώσουμε αυτά τα κενά διαστήματα μεταξύ αυτών των διαδικασιών, δηλαδή να επιταχύνουμε την ανάπτυξη, την, την ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να υλοποιήσουμε ό,τι είναι εφικτό αυτή τη στιγμή. Το απλά να περιμένουμε η ανάκαμψη να φέρει τα αποτελέσματά της χωρίς καμία προσπάθεια δεν επαρκεί. Χρειάζονται ειδικά μέτρα και ειδικά προγράμματα. Έχουμε ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Θέσεων Εργασίας και Απασχόλησης που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και πολλά κράτη-μέλη έχουν λάβει επιπλέον μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Σε γενικέ γραμμέ χρειαζόμαστε περισσότερη διαρθρωτική οικονομική ανάπτυξη πέραν της βραχυπρόθεσμης ε, ε, ανάκαμψης της ανάπτυξης. Το να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μα θα αποτελέσει παράγοντα κλειδί. Η ανταγωνιστικότητά μα δέχεται πολλέ πιέσει, όχι μόνο από τι αναδυνόμενε δυνάμει όπω η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε παρατηρούν τεράστια μείωση ε, των ενεργειακών τιμών χάρη σε νέε ανακαλύψει και βρίσκονται στα πρόθυρα τη επανεκβιομηχάνηση. Γι' αυτό πρέπει ακούραστα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ε, για του ε, παράγοντε κλειδιά της ανταγωνιστικότητάς μας χρησιμοποιώντα τα εργαλεία που επινοήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά πρέπει το φορτίο να μοιράζεται ομοιόμορφα και να διατηρεί την κοινωνική συνοχή. Φυσικά ο απότερος στόχος των προσπαθειών σταθεροποίηση είναι η απασχόληση και η ανάπτυξη. Ε, φύσεως κοινωνικός. Δεν πρέπει ωστόσο ποτέ να χάνουμε από τα μάτια μας τις συγκεκριμένες πολιτικές, ε, κοινωνικές μας πολιτικές. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονό ότι στο Συμβουλίο του Δεκεμβρίου μου ζητήθηκε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνω συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής μας Ένωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, ενώ συνεργαζόμαστε για να ανοικοδομήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα η Ευρωζώνη εμπλέκονται επίσης σε ένα άλλο έργο μεγάλης κλίμακας που συνδέεται στενά με τα προηγούμενα. Είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο, αλλά ήδη αισθανόμαστε τις επιπτώσεις του. Μιλάω για την ενίσχυση της οικονομική και νομισματικής μα ένωσης. Η κρίση μας υπενθύμησε με πολύ σαφή τρόπο ότι η ύπαρξη μιας γνήσιας οικονομικής ένωσης σημαίνει πολλά περισσότερα από το να έχουμε το ίδιο νόμισμα. Το να επιλύσουμε, για να επιλύσουμε τα προβλήματα, το σημερινά οικονομικά προβλήματα, χρειαζόμαστε ένα πιο σταθερό πλαίσιο και πιο σταθερές οικονομικές και νομισματικές πολιτικές. Αυτό το έργο που ξεκίνησε τον Ιούνιο και που αναφέρεται στις τρεις ε, διαδοχές με εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι οποίε ονομάζονται Towards the Genuine Economic and Monetary Union, προ μια γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση, αυτέ οι εκθέσει ε, σημειώνουν πρόοδο βαθμία. Η Τραπεζική Ένωση που μας επέτρεψε να αξιολογήσουμε τους τραπεζικούς κινδύνους καλύτερα και να μειώσουμε το κόστος για τους Ευρωπαίους φορολογουμένους μέσω του ενιαίου ε, μηχανισμού εποπτείας και ενός ε, κοινού μηχανισμού εξυγίανσης έχει φτάσει ήδη σε προχωρημένο στάδιο και το Δεκέμβριο στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, είπαμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών μας πολιτικών ακόμη πιο στενά μέσω εκ των προτέρων συντονισμού των οικονομικών μέτρων στα κράτη-μέλη μας και μέσω συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαρθρωτικές κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Πράγματι, το μεγαλύτερο δίδαγμα που αποκομίσαμε από τα τελευταία χρόνια είναι ο βαθμός τον οποίο είτε μας αρέσει είτε όχι όλοι είμαστε εξαρτημένοι ένας από τον άλλο. Οι αποφάσεις του ενός κράτους μέλους επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό τα τις περιουσίες των άλλων κρατών μελών και τις τύχες των άλλων κρατών μελών στον οικονομικό χώρο, οι τράπεζες σε οποιαδήποτε χώρα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του συνόλου. Η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι είναι η κοινή διαχείριση αυτής της αλληλεξάρτησης και η ανάληψη της κοινή μας ευθύνη. Θέλουμε να διατηρήσουμε στο μέγιστο βαθμό τη δυνατότητα των κρατών μελών να κάνουν τις δικές τους κοινωνικές επιλογές διατηρώντας ένα επίπεδο κοινής ε, χάραξη πολιτική που είναι απαραίτητο για την επιδεύξη των κοινών στόχων. Γι' αυτό το λόγο συναντήσαν αυτή είναι τόσο μεγάλη σημασία. Όπου σε μια κοινή συζήτηση ακούγονται οι εθνικέ ευαισθησίε τη κάθε χώρα μαζί με μια αίσθηση κοινού σκοπού μέσω τη συνεργασία. Είναι θεμελιώδη σημασία για να επιτύχουμε του στόχου μα. Επίση ε, γνωρίζω Έχω απόλυτη αίσθηση ότι υπάρχει ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι όλε μα οι διαδικασίε θα είναι δημοκρατικά υπόλογες και ορατά. Επ' αυτού είναι σημαντικό ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν είναι ανταγωνιστέ. Είναι δύο πλευρέ του ίδιου νομίσματο. Ενώ το καθένα έχει ευθύνε στο δικό του επίπεδο, οι οποίε θα ενισχυθούν, η συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο επίπεδων που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 9 του πρωτοκόλου 1 του Συμφώνου της Λισαβόνας είναι επίσης σημαντικό. Εκ μέρους μου και με βέβαιος ότι το ίδιο ισχύει για τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί σας καθώς καθιερώνετε τις νέες διαδικασίες και μηχανισμούς σας ή ενισχύετε τους υπάρχοντες ώστε να διασφαλίσουμε τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, λογοδοσίας και κοινοβουλευτικής εξέτασης στην ε, βαθύτερη οικονομική και νομισματική μας ένωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλα αυτά καθίστανται ακόμη πιο σημαντικά όταν οι αγορές είναι ήρεμες, διότι σε αυτή την περίπτωση τα θεσμικά όργανα πρέπει να διατηρήσουν την πίεση για οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και για ανάπτυξη και απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αποτελεί εργαλείο κλειδί στη διατήρηση αυτής της πίεσης και σε αυτό το τομέα ο δικός σας ρόλος είναι ζωτικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε του ε, Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ Χέρμαν. Ευχαριστώ το λόγο ο πρόεδρος ε, της Ελλαδικής Βουλής, ο κύριος ε, Πάρετ, παρακαλώ. Πρόεδρε Σούλτς, κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, συγγνώμη, ε, διακεκριμένη κοινοβουλευτική. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στις, στη λήξη της ε, συνδιάσκεψης αυτής για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή οι Ευρωπαίοι και οι Εθνικοί Κοινοβουλευτικοί μπορούν να παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή όταν είπατε ενώπιον του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο, κύριε Σούλτς, ότι υπήρξε μια διάβρωση της κοινοβουλευτικής εποπτείας και αύξηση του διακρατισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα την ιδέα ότι τα κοινοβούλια και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα πλήρη ρόλο στην διαμόρφωση και στην λήψη αποφάσεων σε όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό χαιρετίζω ιδιαίτερα την ιδέα ενός διακοινοβουλευτικού φόρουμ <clears throat> όπως το σημερινό που δίνει σε όλους μας τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό το ότι αυτή η εβδομάδα αυτή η διάσκεψη λαμβάνει χώρα στην αρχή του έτους των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, επίσημη έναρξη του έτους αυτού στην Ιρλανδία. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε και ποια είναι τα ωφέλη που αντλούμε ως Ευρωπαίοι πολίτες στην Ευρώπη. Επιτρέπει επίσης την διοργάνωση συζητήσεων για το τι σημαίνει να είναι κανείς πολίτης αυτής της μεγάλης Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι είναι το μέλλον που θέλουμε να επιτύχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, λόγω της σοβαρής κρίσης που διατρέχουμε αυτή τη στιγμή υπήρξαν υπήρξε πολύ λίγη πολιτική συζήτηση για τα θέματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος όπως παραγωγής χάρη ο ρόλος μας στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Είναι επίσης σημαντικό να μην ξεχάσουμε και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, αλλά και την κατάσταση αυτών στον τρίτο κόσμο που χρειάζονται ακόμα την βοήθειά μας. Πιστεύω λοιπόν ότι σε Ευρωπαϊκό και σε Εθνικό Κοινοβούλιο οι κοινοβουλευτικοί μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για την αποκοινού ανάπτυξη πολιτικών που θα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Εμείς μιλήσαμε και ακούσαμε τους προηγούμενους ομιλητές να αναφέρουν το πρόβλημα της ανεργίας. Στην Ιρλανδία και ξέρω και σε άλλες χώρες είναι παρόμοια η κατάσταση. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανέργων αλλά εξειδικευμένων εργαζομένων που είναι αρχιτέκτονες, είναι ε, μηχανικοί, ειδικευμένα άτομα, τελικά ζουν με επιδόματα ανεργίας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε να χρονίζει. Εμείς ως κοινοβουλευτικοί σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο με το οποίο αυτά τα άτομα μπορούν να λάβουν μέρος σε ενέργειες, σε εγχειρήματα, σε σχέδια στον τρίτο κόσμο και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους και τις δεξιότητές τους για να εκπαιδεύσουν ανθρώπους στον τρίτο κόσμο που μπορούν να βοηθήσουν έτσι να μάθουν οι άνθρωποι αυτοί πώς χτίζουν σχολεία, ε, νοσοκομεία. Να βοηθήσουμε λοιπόν έτσι στον τρίτο κόσμο, αλλά συγχρόνως να καταδείξουμε ότι η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από μόνο μία οικονομική ένωση. Όπως έχει λεχθεί, η μεγαλύτερη μάστιγα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας είναι η ενέργεια των νέων. Είναι κάτι το αφόρητο, δεν μπορεί κανείς να περιμένει το 25% του πληθυσμού να περιδιαβάζει τους δρόμους χωρίς να κάνει τίποτα. Μετά από πολλά χρόνια εκπαίδευσης σχολικής και πανεπιστημιακής να είναι άνεργοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να βρούμε λοιπόν και πάλι τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βρούμε νέους τρόπους να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό μαζί με τους εταίρους μας. Θεωρώ επίση ότι αξίζει τον κόπο να σας ενημερώσω και για την κατάσταση της οικονομίας της Ιρλανδία και την κατεύθυνση που ακολουθεί. Να σας πω ότι πολλοί είχαν αμφιβολίες για την αξία της ε, συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του είπα δεν ξέρετε ποιοι είναι οι φίλοι σα μέχρι να τους χρειαστείτε. Μας βοήθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ήμασταν σε δύσκολη κατάσταση. Έχουμε αναπτύξει προβλήμα, προγράμματα εθνικής σταθερότητας και μεταρρύθμισης. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντική άσκηση. Ήταν δύσκολη η μεταρρύθμιση. Μετά από όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα μειωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά 12% κατά 37.500 και θα υπάρξουν επίσης περικοπές σε μισθούς, σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς και ιδίως στους πολιτικούς θα υπάρξει συρρήκνωση υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και θα διευρυνθεί η φορολογική βάση με νέους φόρους ακινήτου περιουσίας. Το ανώτατο επίπεδο φορολογίας ήταν 43,5% το 2008 και ξεκινούσε σε εισόδημα 100.000 ευρώ και άνω. Το 2012 μετά από τέσσερα χρόνια το ανώτατο ποσοστό φορολογίας φτάνει το 52% και ξεκινάει στις 32.800 ευρώ. Αυτά δείχνουν τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν στον τομέα της ε, φορολογίας και της, των κοινωνικών παραχών. Εμείς προσπαθήσαμε λοιπόν να μην επιφέρουμε φόρους οι οποίοι θα θίξουν την ανταγωνιστικότητα και το ε, μοναδίο εργασιακό μας κόστος έχει μειωθεί και επομένως αυξήθηκε και η ανταγωνιστικότητά μας όπως φαίνεται και από τι εξαγωγέ μας που αυξάνονται. Όλα αυτά έγιναν με την υποστήριξη των εταίρων μας τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά ξεκίνησαν από εσωτερικές αποφάσεις και βασίστηκαν και στην ανθεκτικότητα και αντοχή του λαού τη Ιλλανδίας. Είναι μια ευαίσθητη ισορροπία η οποία πρέπει να προστατευτεί για το μέλλον. Θα πρέπει να έχουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων κοινοβουλίων για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια ευνοϊκή λύση στα προβλήματα <coughs> χρέους της Ιρλανδίας και θα υπάρξει μια πλήρης εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2012 Θέλω να σας υπενθυμίσω και πάλι τα πολύ θερμά λόγια του Πρόεδρου Σούλτς όταν μίλησε ενώπιον τη Βουλή μα τον Οκτώβριο του 2012, τον παραθέτω. Όταν ένα μέλο τη οικογένεια έχει προβλήματα, τα άλλα μέλη τη οικογένεια θα πρέπει να τον αρρωγήσουν. Είναι στο συμφέρον όλοι μα, η Ιρλανδία να βγει από το μνημόνιό τη το ταχύτερο δυνατό και ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί χάρη στα μέτρα τα οποία ακολουθούμε, αλλά και με τη βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων μας. Τα τελευταία χρόνια περάσαμε μεγάλες δυσκολίες για τα θέματα της οικονομικής διακυβέρνησης. Τραπεζική κρίση, κρίση κρατικού χρέους, ανάπτυξης και ανεργίας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Μας λέγανε κάθε μέρα ότι το ευρώ θα καταρρεύσει, ότι θα επιβιώσει, ότι υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να διασπαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτο σέλιδα άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες κάθε μέρα για την καταστροφή που θα οδηγούσε μετά από αυτή τη διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά βρισκόμαστε τώρα στο 2013, το ευρώ εξακολουθεί να υπάρχει και ενισχύεται κάθε μέρα, οι τράπεζες αναδιαθρώνονται, μειώνονται τα ελλείμματα, βέβαια έχουμε πολύ δρόμο να διατρέξουμε, έχουμε ακόμα 27 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και άλλα κράτη τα οποία θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό είναι ένας φόρος τιμής προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι μεν αισιόδοξο, αλλά δεν θέλω να παραγνωρίσω τις δυσκολίες και τις αδυναμίες που παραμένουν. Πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα του ελλείμματος επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ των Ευρωπαίων, Ευρωπαίων ηγετών και των πολιτών τους για τα ευρωπαϊκά θέματα. Δυστυχώς μιλάμε ε, μόνο αρνητικά συνήθως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν εφαρμόζονται νέοι κανόνες και νέες διατάξεις που ουσιαστικά αποτελούν κυρώσεις προς μερικά κράτη-μέλη. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο και να επικοινωνούμε πιο ανοιχτά με τους πολίτες για τα θετικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα απόσπαστο τμήμα των προσπαθειών που θα πρέπει να καταβάλουμε τα επόμενα χρόνια μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Είμαι 40 χρόνια στην δημόσια ζωή, στην πολιτική ζωή. Μπήκα στην πολιτική λίγο μετά από την είσοδο της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1973. Και μπορώ να θυμηθώ την εποχή αυτή που υπήρχε ακόμα ένα πολύ ψηλό επίπεδο καχυποψίας, ζήλιας, φόβου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πάρει τι αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων και θα συμβούν τόσο τόσα πολλά τρομερά πράγματα. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Με τα χρόνια ο κόσμος έχει κατανοήσει καλύτερα ότι η συνεργασία των κοινοβουλίων μπορεί να οδηγήσει σε πολυθετικά αποτελέσματα και ελπίζω πράγματι ότι αντιμετωπίζοντας το θέμα της επικοινωνίας θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την επικοινωνία με τους πολίτες όλοι από κοινού. Ως παράδειγμα, όλοι μας προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε το ότι θα υπάρχουν κοινοβουλευτικά κανάλια τηλεόρασης. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει ένα κανάλι όπου θα μπορεί κανείς να βλέπει τις ε, ολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις συνεδριάσεις των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να είναι προσβάσιμες σε όλους οι συνεδριάσεις της Κομισιόν και του Συμβουλίου στην κοινοβουλευτική αυτή τηλεόραση. Θα ήθελα να βλέπω επίσης και να υπάρχει δυνατότητα των Ιλλανδών και άλλων Ευρωπαίων να παρακολουθούν τα τεκτενόμενα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει την αντίληψη που έχουν οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάποιο βαθμό όλη η πολιτική είναι τοπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τα ευρωπαϊκά θέματα να έχουν <clears throat> ορατότητα και σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό εγώ προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μου με τους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν και σε όλες τις πτυχέ ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τους πολίτες και την μείωση του ελλείμματος επικοινωνίας και θέλω να ευχηθώ σε όλους αυτούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα αντιμετωπίσουν την εκλογική διαδικασία του χρόνου. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να λάβω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε Μπάρετ. Λοιπόν, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει ένας πολύ ε, γνωστός Γερμανός ε, ηθοποιός και κομικός, ο Καρλ Βάλεντιν, και είχε πάει στη Βαβαρική Βουλή κάποια φορά και είπε Τώρα καταλαβαίνω τι είστε κοινοβουλευτισμό. Υπόθηκαν τα πάντα, αλλά όχι ακόμα από όλους. Και γι' αυτό το λόγο ε, δεν θα βγάλω κι εγώ τώρα λόγο, διότι έχω καλυφθεί από όλους τους προλαλήσαντες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον πρόεδρο του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου που μύρισε ε, πραγματικά από την καρδιά του και εξέφρασε και αυτά που πιστεύουμε εμείς. Έχουμε ε, το Europal TV που είναι το κανάλι της τηλεόρασης και μπορούμε πολύ εύκολα να δικτυωθούμε με εθνικά κανάλια. Και αν αρχίσει η Ιρλανδία θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Είναι βέβαιο αυτό. Σας προτείνω τώρα να μπείτε και εσείς στη συζήτηση, την οποία θα προεδρεύσει η συνάδελφος Άννη Ποδηματά. Ζητώ συγγνώμη γιατί σε λίγο έχω μια συνάντηση, θα υποδεχτώ τον ε, Πρωθυπουργό της Λιθουανίας και αμέσως μετά ε, τον ε, Πρωθυπουργό το τοπικό και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας. Έχω πολύ σημαντικά καθήκοντα παραστάσεις τώρα, αλλά δεν θέλω να φύγω χωρίς να σας πω κάτι προσωπικό. Πέρα από ε, τις πολλές και μεγάλες ευχαριστίες που θα ήθελα να σας απευθύνω για την παρουσία σας, θα ήθελα να σας θυμίσω τη σημερινή ημερομηνία. Σήμερα έχουμε 30 Ιανουαρίου. Πριν από 80 χρόνια ακριβώς, άρχισε η πιο σκοτεινή περίοδος της ιστορίας της Υπήρου μας. Στις 30 Ιανουαρίου του 1933, ο εγκληματίας αυτός της ανθρωπότητας, ο Αδόλφος Χίτλερ, άρπαξε την εξουσία στη Γερμανία. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν αυτή την ημέρα, τα πρώτα 12 χρόνια της ζωής τους, έζησαν φρίκη, καταστροφή, διάλυση, εξολόθρευση, ε, αφανισμό. 80 χρόνια αργότερα, σήμερα, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση είμαστε εδώ ευρωβουλευτές και βουλευτές Εθνικών Κοινοβουλίων 27 κρατών μελών. Όλων των εθνών, όλων των φυλών, όλων των θρησκειών, όλων των απόψεων. Όλοι αυτοί εκπροσωπούνται από κοινού εδώ για να συζητήσουμε για το μέλλον των παιδιών που γεννιούνται σήμερα. Και ε, Μάλιστα από κοινού όχι ο ένας απέναντι στον άλλον μια μέρα σαν τη σημερινή θα πρέπει να σκεφτούμε τι συναρπαστική ιστορική πρόοδος είναι αυτή η δυνατότητα που έχουμε σήμερα να το πράττουμε αυτό. Γι' αυτό είναι τόσο αντιπροσωπευτική η σημερινή αυτή η συνεδρίαση. Το ευρωπαϊκό πνεύμα που εκπροσωπούμε όλοι μας. Είτε λειτουργούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εργαζόμαστε είτε σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το πνεύμα λοιπόν είναι το καλύτερο μέσο για να αποτρέψουμε τέτοιου είδους εγκληματίες που ανέλαβαν την εξουσία τότε στη Γερμανία ε, που ε, έβαλαν φωτιά και στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο. Να αποφύγουμε λοιπόν να επανέλθουν τέτοια φαινόμενα. Η εργασία μας θα πρέπει να συνεχιστεί και υπό αυτό το πρίσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από όλα αυτά τα λόγια που ακούσαμε υπέρ του κοινοβουλευτισμού, αυτά τα όμορφα λόγια, εμείς τα μέλη των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και τις δύο προηγούμενες μέρες, χθες και προχθές, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε και να αποδείξουμε την τεράστια αξία του κοινοβουλευτισμού που όπως ε, υπογράμμισαν όλοι οι αξιότιμοι ομιλητές ε, αντιπροσωπεύει τεράστια αξία και διατρέχει τεράστιο κίνδυνο σήμερα. Ανοίγω λοιπόν τη συζήτηση, απλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχετε κάρτες ομιλίας ε, στα γραφεία σας με τις οποίες μπορείτε να μας υποδείξετε ότι θέλετε να λάβετε το λόγο. Εφόσον το επιθυμείτε, παρακαλώ, συμπληρώστε μια τέτοια κάρτα και διαβιβάστε την σε εμάς. Αυτό ισχύει στα, τόσο για τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων όσο και για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο χρόνος ομιλίας θα περιορίζεται σε τρία λεπτά και ίσως χρειαστεί να τον αναπροσαρμόσουμε. Εάν δούμε ότι ο χρόνος εξαντλείται θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία με χθες. Αυτό σημαίνει ότι δύο εθνικοί βουλευτέ θα λαμβάνουν το λόγο και μετά ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανοίγω λοιπόν τη συζήτηση και δίνω το λόγο πρώτα στην κυρία Χέλγα που είναι πρόσωπος της Επιτροπής Προπολογισμού στη Γερμανία. Έχετε το λόγο. Όχι, είμαι μέλος όμως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη Γερμανία. Είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ίσως να μιλήσουν πρώτα δύο εκπρόσωποι εθνικών κοινοβουλίων. Συγγνώμη, υπήρξε μια σύγχυση εδώ με τις κάρτες. Η κυρία Μπετίνα Κούντλα, λοιπόν, από τη Γερμανία έχει πρώτη το λόγο. Παρακαλώ, για τρία λεπτά. Μπετίνα Κούντλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι ήταν σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε συγκεντρωθεί εδώ στη διακοινοβουλευτική διάσκεψη, η οποία τόνισε και πάλι και κατέδειξε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση που να επιτρέπεται να λαμβάνεται ερήμην του λαού, χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση. Το θέμα αυτό αναφέρθηκε και ακούσαμε ότι ενδεχομένως η Μεγάλη Βρετανία να κάνει δημοψήφισμα. Και τη με. Γιατί φοβόμαστε γενικά τα δημοψηφίσματα. Κανονικά θα πρέπει να τα καλωσορίζουμε και μόνο. Εάν μπορούμε να αναμένουμε ότι σε όλα τα κράτη ε, ο πληθυσμός εκφράζεται φιλοευρωπαϊκά και λαμβάνει ε, ξεκάθαρη θέση. θα πρέπει να φοβόμαστε τα δημοψηφίσματα μόνο σε περίπτωση που ε, υπάρχει φοβός για αρνητική έκβαση και που φοβούνται οι πολίτες ότι δεν ε, ακούγονται τα μελήματά τους και δεν έχουν καμία δυνατότητα μέσω των εθνικών τους κοινοβουλίων να επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες. Σύντομα θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια θέματα ε, ουσιαστικά που ακούσαμε τις περασμένες μέρες. Ο κύριος Μπαρόσο τονίζει πάντα την έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Για το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο ε, θα πρέπει λέει, να έχουμε υπόψη μας και να φέρουμε στο προσκήνιο αυτό το θέμα της προστιθέμενης αξίας. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα εφιστάμενα πλαίσια τις δαπάνες ε, που τρέχουν ε, με βάση τις ηλμένες αποφάσεις. Αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν γιατί παραμένουν 250 δισεκατομμύρια ε, ευρώ υπόλοιπα του προϋπολογισμού, δηλαδή από έργα, από τον τρέχοντα προϋπολογισμό που δεν έχουν ακόμα δεσμευθεί. Λοιπόν, ας απορροφήσουμε πρώτα αυτά τα κονδύλια πριν μπούμε σε νέες οικονομικές απαιτήσεις και δημοσιονομικές για το θέμα της ε, εγγύησης για τους νέους. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης. Καλωσόρισε ρητά ε, τη δυνατότητα αυτή για τις μεμονωμένες κυβερνήσεις και τη μεγαλύτερη προσήλωση των κυβερνήσεων εκεί. Η νεολαία θα πρέπει να έχει προοπτική εντός της Ευρώπης. Ταυτόχρονα όμως τέτοιες εγγύησεις θα πρέπει να είναι αμυγός εθνική υπόθεση. Μπορεί σε ορισμένες χώρες όπως είναι η Φιλανδία ε, να υπάρχει δυνατότητα να δοθεί μια τέτοια εγγύηση. Θα πρέπει όμως να αναλύσουμε αν κρατικές εγγύησεις είναι μάλλον βάρος και μεγάλο για τα κράτη με τόσο μεγάλη ανεργία νέων. Δηλαδή να υπόσχονται κάποια πράγματα τα κράτη που δεν θα είναι σε θέση στη συνέχεια να τα τηρήσουν. Και το μέγα πρόβλημα της ανεργία των νέων δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τα πλαίσια για να αναπτυχθεί, για να ξεδιπλωθεί ιδιωτική πρωτοβουλία και να δημιουργήσουν θέσει εργασία επιχειρήσει. Δεν μπορεί το κράτο από μόνο του να υπομειστεί τέτοιο βάρο. Κοινωνικό είναι αυτό που δημιουργεί θέσει εργασία. Κοιτάξτε και την ώρα, λέει η πρόεδρο. Να δεν βλέπω ρολόι εδώ. Ε, ναι, έχετε δίκιο. Το βάλαμε μπρο το ρολόι με καθυστέρηση, αλλά έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Μάλιστα. Τελειώνω λοιπόν. Και συνοψίζω. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνουμε στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την εποπτεία των τραπεζών και για το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Γιατί με ενόχλησε κάπως το γεγονός ότι από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται λόγος μόνο για την Τραπεζική Ένωση και όχι για την Τραπεζική Εποπτεία. Οι αποφάσεις που παίρνει το δικό μας κοινοβούλιο λέγουν ότι η Γερμανική Βουλή Bundestag συμφωνεί για τράπεζες ε, που έχουν σημασία συστημική θα πρέπει να υπάρχει μια τραπεζική εποπτεία, αλλά ε, απορρίπτουμε την Τραπεζική Ένωση που σημαίνει κοινοτικοποίηση και συνένωση των καταθέσεων. Κάτι τέτοιο δεν στερείται δημοκρατικής νομιμότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να ρωτήσω αν έχει ρυθμιστεί το ρολόι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, διότι οι ομιλητές χρειάζεται να τηρούν το χρονομιλία τους. Okay, then I will now give... Ωραία, λοιπόν, δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Οίκο που είναι γραμματέα Ευρωπα... της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Λετωνία. Okay. Yes, uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα λετωνικά. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο από το 2014 μέχρι το 2014 είναι πολύ σημαντικό για τη Λετωνία. Είναι πολύ σημαντική η διαμόρφωσή του για τη Λετωνία, διότι η οικονομία μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κονδυλία αυτού του ε, προϋπολογισμού. Το επόμενο δημοσιονομικό, ε, το, ο επόμενος ετήσιος προϋπολογισμός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο των συζητήσεων. Στο μεταξύ χρειαζόμαστε να δούμε τι θα γίνει με τα, ε, ταμεία συνοχής. 1,5% του ΕΠ αντιστοιχούν αυτά. Στο μεταξύ φαίνεται ότι ότι η χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχή θα μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και αυτό θα εξαρτηθεί από τι μακροοικονομικέ πρόβλεψει και θα μπορούσε να πω 0,6 έω 1 δι ευρώ. Η νέα προγραμματική περίοδος για την περίοδο συνοχής ε, για τις χώρες έχει μειωμένα ανώτατα επίπεδα τα οποία έχουν υπολογιστεί βάσει των προηγούμενων δικτών ΑΕΠ. Αυτό επηρεάζει αρνητικά το κονδύλιο για την Λετωνία, διότι στην αρχή της κρίσης η Λετωνία υπέστη πολύ γρήγορη ύφεση και συνεπώς οι μακροοικονομικοί δείκτες εκείνη τη στιγμή υποβαθμίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Στο Λετωνικό Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν διάφορα επίπεδα πιστώσεων για τις χώρες εκείνες που στην περίοδο 2008-2010 ε, είχαν πολύ χαμηλή ανάπτυξη του ΑΕΠ, πολύ πιο ε, χαμηλή ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, όταν αυτές οι χώρες έχουν πολύ, καλούς, πολύ καλά ποσοστά απορρόφησης, τότε η χρηματοδότηση συνοχής θα πρέπει να διασφαλίζεται σε τέτοια επίπεδα που να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020. Τώρα, μιλώντας για την κοινή γεωργική πολιτική, η μέση άμεση ενίσχυση στη Λετωνία ήταν η χαμηλότερη, το χαμηλότερο ποσό από όλα τα κράτη-μέλη, 34% μόλις του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο άμεσης ενίσχυσης το μέσο ποσό, ο μέσος όρος των άμεσων ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν πιο δίκαιο. Ε, καλό θα ήταν ε, να φτάνει τουλάχιστον το 80% του μέσου όρου. Αυτή δεν θα έπρεπε να μειωθούν η χρηματοδότηση για την γεωργική ανάπτυξη ή για την αλληλεία Τονίζω ότι χαμηλότερα επίπεδα αναπτυξιακής χρηματοδότησης υποβαθμίζει την κατάσταση χωρών που αρχίζουν να εξέρχονται από την κρίση και μειώνει την ανταγωνιστικότητά τους. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρος. Τώρα κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να τονίσω δύο βασικές ιδέες που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Η πρώτη ήταν η δέσμευση του Προέδρου κ. Παρόσο ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία, μάλλον δήλωση, αποδεικνύεται από την ενίσχυση ε, του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων απέναντι στο Συμβούλιο. Σωστή είναι αυτή η δήλωση. Και αυτό τι σημαίνει. Ότι και εμείς εδώ, αλλά και εσείς ε, στις χώρες σας, θα πρέπει να έχουμε την αξίωση να συνεργαζόμαστε στενά για να μπορέσουμε να διαδραματίσουμε το ρόλο μας απέναντι στο Συμβούλιο, να του δίνουμε εντολές, να το ελέγχουμε, αλλά να είμαστε σε ένα γνήσιο διάλογο. Ε, εμείς ε, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παρατήρηση δεύτερη που θεωρώ πολύ σημαντική για σήμερα. Στους Financial Times βλέπουμε και διαβάζουμε ότι οι 11 χώρες που θέλουν να εισαγάγουν το φόρο χρηματοπιστωτικό συναλλαγών υπολογίζεται ότι τα ε, έσοδά τους θα είναι 30 με 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθόλου ευκαταφρόνει το πόσο. Γνωρίζετε ότι κάνουμε τώρα τις διαπραγματεύσεις ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν έχουμε τέτοια έσοδα που είναι το 1 τέταρτο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι πολύ σημαντική συνεισφορά. Το αναφέρω τώρα εδώ διότι με τα κράτη-μέλη υπάρχει ένας τεράστιος καυγάς ακόμα για το πού θα πάνε τα λεφτά αυτά και ποιος θα τα συλλέγει και ποιος θα τα αξιοποιεί. Ε, τα κράτη-μέλη ε, έχουν την αξίωση να πάνε στα εθνικά κοινοβούλια, ενώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συντριπτική η πλειοψηφία που λέγει ότι είναι πολύ σημαντικό τα έσοδα αυτά να γίνουν ίδιο πόρος του κοινοτικού προπολογισμού και με τον αντίστοιχο τρόπο ε, οι συνεισφορές των κρατών του ΑΕΠ τους δηλαδή, να μειωθούν των κρατών που είναι πρόθυμα να υιοθετήσουν το φόρο αυτό. Σε καιρούς κρίσης λοιπόν απαντούμε έτσι και σε περίοδους εξυγίανσης ε, των ε, κρατικών και εθνικών προϋπολογισμών έχουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα πού θα βρούμε χρήματα για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ιδού, ξέρω ότι είναι πολύ επίμαχο σε πολλά κράτη και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλανδία και αλλού αλλά σας παρακαλώ να ε, το σκεφτείτε αυτό, γιατί έχουμε την έκτακτη σύνοδο κορυφή την άλλη εβδομάδα και θα τους απασχολήσει και αυτό, όπως και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να αποφανθούν και θα είναι αποφασιστικό για το μέλλον του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τρούπελ και ευχαριστούμε για την αναφορά στο φόρο περί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Σέρβέ από τι κατοχώρε. Yes, uh, thank you, Chair. Um, let me uh, Ξεκινώ λέγον ότι νιώσαμε κάποια απογοήτευση για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Κομισιόν αλλά και ο πρόεδρος του Συμβουλίου αναγκάστηκαν να φύγουν μετά την ομιλία τους. Θα θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί τους. Δεν αρκεί να λέμε ότι τα, ευρωπαϊκά, τα εθνικά κοινοβούλια σημαντικά, θα πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί τους. Βλέπω όμως ότι ο Επίτροπος κ. Σεύκοβιτς είναι παρόν ακόμα και παίρνω την ευκαιρία να του θέσω ένα ερώτημα. Τις δύο τελευταίες μέρες συζητήσαμε για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στον κοινοβουλευτικό έλεγχο των κυβερνήσεών τους και μιλήσαμε και για την δημοκρατική νομιμοποίηση και τη διαφάνεια. Για τη διαφάνεια. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Είχαμε πολλές διασκέψεις κορυφή τα τελευταία χρόνια με απόλυτα αδιαφανή προετοιμασία. Αν δούμε παραδείγματο χάρη το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, μία εβδομάδα πριν από το Συμβούλιο παρουσιάστηκε η πρόταση της Κομισιόν από τον κύριο Μπαρός. Και λίγες μέρες πιο πριν από την διάσκεψη κορυφής εμφανίστηκε το έγγραφο Φαν Ρομπάι. Για μας ήταν αδύνατο στο Κοινοβούλιο να έχουμε μια πλήρη συζήτηση για τα έγγραφα αυτά. Και τα σχέδια απόφασης των Ευρωπαϊκών συμβουλίων δεν είναι διαθέσιμα για τους απλούς πολίτες. Είναι περιορισμένου χαρακτήρα έγγραφα. Καμιά φορά μπορούμε να τα διαβάσουμε, αλλά δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτά σε συζητήσεις και δεν είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό. Το ερώτημα μου προς την Κομισιόν είναι λοιπόν πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Λήψης Αποφάσεων και κατά πόσο θα ήταν υπέρμαχος όπως εμείς του να γίνουν τα έγγραφα του Συμβουλίου ανοιχτά και στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρύ Κοινό. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Δεκρούφ από το Βέλιο. Εκτός μικροφώνου μιλητής. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ακολουθούμε και παρακολουθούμε τη συζήτηση και βλέπουμε ότι το, πρόγραμμα της, ε, το πρόβλημα συγγνώμη, δημοκρατικής νομιμοποίησης είναι πάρα πολύ έντονο. Ποιοι όμως υπερασπίζονται τη δημοκρατική νομιμότητα. Λένε ναι μεν αλλά. Γιατί όταν κάποιος επιθυμεί να είναι ένθερμος και διάπειρος ε, υποστηρικτής ε, ενός θέματος στερείται νομιμότητας. Γίνεται αυτή η συζήτηση όλο και περισσότερο. Ποια είναι η νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι εκλεγμένο, με δημοκρατικό τρόπο, ε, λειτουργεί δημοκρατικά και δραστηριοποιείται, αλλά στην ουσία όπου έχει συναπόφαση ε, αυτό αφορά το 1% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Από την άλλη έχετε στις 27 χώρες 40 κοινοβούλια. Κάθε χρόνο ανανεώνονται 4 με 5 κοινοβούλια και έχουν λόγο τεράστιο για 50% περίπου του ΑΕΠ της χώρας τους εκάστοτε. Έχω την τιμή ή βρίσκομαι στην κατάσταση να έχω διατελέσει πάνω από 45 χρόνια εκλεγμένος βουλευτής σε μια Εθνική Βουλή και μάλιστα είχα την ευκαιρία να διατελέσω και πρόεδρος της Βουλής και διαπίστωσα πόσο δύσκολα ε, η ευρωπαϊκή ε, πολιτική βρίσκει το δρόμο της στα εθνικά κοινοβούλια. Οχτώ χρόνια ήμουν πρόεδρος ε, πριν από το Χέρμαν Φαν Ρομπάι της Βολής των Αντιπροσώπων στο Βέλγιο και σε όλους τους κανονισμούς που ήμασταν υποχρεωμένοι να συζητάμε προσπαθούσαμε ε, κάθε φορά να το βάζουμε στην ημερήσια διάταξη των επιτροπών και δεν είχε τρελαθεί ο κόσμο από ενθουσιασμό. Με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια και του τελευταίους μήνε συγκεκριμένα. Γιατί εδώ μπαίνει πολύ βαθιά η Ευρώπη στα πράγματα στην Ευρωζώνη με ε, τις παρεμβάσεις και επεμβάσεις στους προϋπολογισμούς, ε, με όπου γίνεται εξίσωση της οικονομικής, κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής και καταλαβαίνει ο κόσμος ότι επεμβαίνει η Ευρώπη στη ζωή του, όχι με κανόνες για ε, διευκόλυνση και απλούστευση της ε, ελεύθερης αγοράς, αλλά και για θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Και εγώ προβληματίζομαι και διαρωτώμαι και τελειώνω με αυτό. Επικορικότητα ακούμε, αναλογικότητα ακούμε. Μα αυτό αν το επεκτείνουμε σε μεγάλα προβλήματα, ε, έχει δικαίωμα η Ευρώπη να αναμειγνύεται σε αυτά. Δεν ξέρω, μήπως χρειάζονται συμφωνίες περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεκρό. Αγαπητοί συναδέλφοι, ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι ο κύριο Μπαρόζο, ότι ο πρόεδρο Μπαρόζο έφυγε, όπω γνωρίζετε, αλλά ο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Σεύκοβιτ, βρίσκεται μαζί μα. Αφού ολοκληρωθεί αυτός ο πρώτος ε, γύρος ομιλιών, θα του δώσουμε το λόγο και πιθανώς επειδή έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας, ε, θα έχετε την ευκαιρία, τη δυνατότητα να του υποβάλλετε κάποιες ερωτήσεις και σε δεύτερο γύρο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον διάδελφο Χουαγκό. Ευχαριστώ πολύ Άννη. Δεν ήθελα απαραίτητα να μιλήσω διότι μίλησα χθε ε, για την ετήσια επισκόψη της ανάπτυξης που μου φαίνεται η συζήτηση κλειδί αυτή τη στιγμή σε αυτό το ευρωπαϊκό εξάμενο αλλά δυστυχώς δεν είναι νομοθετική πράξη. Εδώ απλά μιλάμε για διάφορα αλλά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ήθελα απλά να αντιδράσω στα όσα είπε ο συναδέλφος ε, του Γερμανικού Κοινοβουλίου που κατήγγειλε τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της Τραπεζικής Ένωσης. Θα ήθελα να του υπενθυμίσω ότι η Γερμανίδα Καγκελάριος ήταν αυτή που πρότεινε αυτή την Τραπεζική Ένωση ως ε, αντίτιμο για την επακεναφαλοποίηση των Ισπανικών τραπεζών και αυτό μας βοηθάει να αποφύγουμε μάλλον μια δεύτερη εξαιρετικά ε, ε, δυνατή τραπεζική κρίση στην Ευρώπη. Η Τραπεζική Ένωση σήμερα πρέπει να περάσει, θα αποτελέσει άλλο ένα βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η Γερμανία από αυτή την άποψη ε, διδασκεί ολόκληρη την Ευρώπη ε, μας ζητάει να προχωρήσουμε σε αυτή την ομοσπονδία και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ομάδα των Σοσιαλιστών ιδιαίτερα είμαστε υπέρ σε μεγάλο μέρος ε, αυτής της ομοσπονδίας αλλά το θέμα είναι να είναι δημοκρατική Τα ωραία λόγια δεν ε, χρησιμεύουν. Τα εθνικά κοινοβούλια φυσικά θα πρέπει να παίζουν το ρόλο τους ε, στις χώρες τους, να εποπτεύουν ε, τις χώρες τους με δημοκρατικό έλεγχο, αλλά σε ευρωπαϊκή κλίμακα έχουμε επίση ένα δημοκρατικό διακύβευμα. Και εμείς θα θέλαμε αυτή η τραπεζική ένωση να ελέγχεται δημοκρατικά. Γι' αυτό το λόγο στην έκθεση της ζητήσαμε ρητά και το Κοινοβούλιο το υπερψήφισε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας να αποτελεί το αντικείμενο δημοκρατικής διακυβέρνησης και όχι απλά να είναι διακυβερνητικός. Πολλά τέτοια λοιπόν δημοκρατικά εργοτάξια στα οποία πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι με από κοινού κυριαρχία μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού κοινοβούλου, αντί να ερχόμαστε ένα αντίθεση με τον άλλο. Merci. Ε, Ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον γερουσιαστή Τέρι Λέιντεν από την Ιρλανδία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που βρίσκομαι εδώ με τα μέλη των κοινοβουλίων 27 χωρών και τους ευρωβουλευτές και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου που συνέβαλε ιδιαίτερα στη σημερινή συζήτηση. Δεν έχει πολλές ευκαιρίες ε, να εκφράσει τις απόψεις του για διάφορα ζητήματα και και ιδιαίτερα που τις άκουσα. Ε, είναι πολύ σημαντικό που μοιράστηκε τις απόψεις του εδώ. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η οι προτάσεις που υπέβαλε, οι συστάσεις του, η κινητοποίηση των εργαζομένων που έχουμε μηχανικών και των εξειδικευμένων εργαζομένων. Όλα αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ιρλανδία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργαζόμενοι όσοι είναι άνεργοι θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν, να απασχοληθούν χρήσιμα στο να χτίσουν σχολεία και κατοικίες και νοσοκομεία. Όπως γίνεται σε μια αντίστοιχη περίπτωση στην Νότια Αφρική, ε, Είναι μια εξαιρετική πρόταση που υποστηρίζω απόλυτα. Επίσης όσον αφορά την κάλυψη των ευρωπαϊκών υποθέσεων, την ε, ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη των υποθέσεων των εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Ε, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, αλλά δεν υπάρχει αρκετή κάλυψη. Υπάρχει κάποια κάλυψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αργά το βράδυ. Πιστεύω θα άξιζε τον κόπο να το υποστηρίξουμε αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να το υποστηρίξει. 40 χρόνια βρίσκεται η Ιρλανδία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ, στην τότε ΕΟΚ. Ήταν εξαιρετική εμπειρία. Αναμφίβολα ο λαός της Ιρλανδίας έχει επικυρώσει όλα τα δημοψηφίσματα σε σχέση με τις αλλαγές και τις συνθήκες σε όλο αυτό το διάστημα. Πίστευουμε ότι πραγματικά άξιζε τον κόπο όταν, συναντάμε, όταν συναντήσαμε μεγάλες δυσκολίες πριν από 3-4 χρόνια υπήρξε τεράστια υποστήριξη προ την Ιρλανδία αλλά το κόστο αυτή τη υποστήριξη είναι εξαιρετικά βαρύ αυτή τη στιγμή ε, αφορά το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλα αυτά τα χρέη είναι οπωσδήποτε είναι ζωτική σημασία να το επαναδιαπραγματευτούμε. Όλο αυτό οι Ιρλανδοί έχουν υποφέρει. Εμείς υποστηρίξαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν και την Ευρωζώνη. Και χωρίς αυτές τις αποφάσεις του της Ιρλανδικής κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων πιστεύω ότι θα είχε υπάρξει τεράστια κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Ήθελα να συγχαρώ και τους συναδέλφους μου για τις συμβολές τους και τα μέλη των αντιπροσωπείων εδώ. Πραγματικά άξιζε αυτή η άσκηση από τη δική μου άποψη ως μέλος της Ιρλανδικής Γερουσίας και μέλος του ε, Συμβουλίου της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γερουσιαστή Λέιντεν. Να έχετε δίκιο. Πράγματι έχει συμβάλει εξαιρετικά το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο σε αυτές τις δύο ημέρες συζητήσεων, ειδικότερα φυσικά ο εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου. Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ε, έχω άλλο ένα αίτημα από τον κύριο Σαλαβράκο, τον οποίο δεν βλέπω εδώ στην αίθουσα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαρος για ένα πρώτο γύρο απαντήσεων στα όσα είπατε και όσα ρωτήσατε. Και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους προέδρου, στην Πρόεδρο της ε, Επιτροπής ε, Απασχόληση ε, και Προπολογισμού, την κυρία ε, Μπερέ και τον κύριο Λαμασούρ, που θα ήθελα να σχολιάσουν τι ομιλίε που άκουσαν μέχρι στιγμή. Στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία, σα υπενθυμίζω ότι έχετε αυτέ τι κίτρινε κάρτε στα γραφεία σα, να ζητήσετε τον λόγο. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση περίπου στι 12, 12 και 4. Κύριε Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ για την ευκαιρία να απαντήσω στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Θα προσπαθήσω να τι απαντήσω στη σειρά που ετέθηκαν. Η κυρία από την, ε, από την ε, Γερμανική Bundestag μας υπενθύμησε ότι πρέπει να δίνουμε περισσότερη έμφαση στην προσθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και συμφωνώ γιατί όπω είπε και ο πρόεδρος τη Επιτροπή. Πολλέ φορέ στη συζήτηση που γίνεται για τι δημοσιονομικέ πρόπτικες λησμονούμε Είμαστε επιλύσμονες του γεγονότος ότι η συμφωνία για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές ωφελεί όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και τα οποία αναφέρθηκαν και στη συζήτηση η οποία λαμβάνει χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ελπίζω ότι θα είναι και στοιχεία της συνεχιζόμενης αυτής της συζήτησης. δείτε τα πρόσφατα στοιχεία, η συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου το 2011 ήταν περίπου 6 δισεκατομμύρια λίρες, περίπου 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και οι εκτιμήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ότι το, τα αιτήσια ωφέλη για τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και τους πολίτες είναι 30 με 90 ε, δισεκατομμύρια λίρες. Αυτό εξαρτάται βέβαια από τη φάση του οικονομικού κύκλου. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δει κανεί με αυτόν τον τρόπο τον ευρωπαϊκό προπολογισμό ότι δεν είναι μονάχα το 1% του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το συνολικό όφελο το οποίο προσποριζόνται τα κράτη-μέλη. Όταν ήμουνα στι κάτω χώρε, συζητούσαμε τι συνέπειε τη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και ένιωσα μεγάλη χαρά όταν το Γραφείο σχεδίαση των Κάτω Χωρών επιβεβαίωσε ποια είναι τα ωφέλη για τους Ολλανδούς πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 2.000 ευρώ κατά κεφαλή το χρόνο ήταν το όφελος. 7 με 8 φορές δηλαδή περισσότερο κατά κεφαλή από ότι είναι η καθαρή συνεισφορά της Ολλανδίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά για να γίνει κατανοητό ότι μέσα από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την ενία αγορά, μπορούμε να έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις και τους πολιτές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν θα πρέπει να βλέπουμε μια στενόμια λογιστική με μια στενόμια λογιστική αντιμετώπιση τον προπολογισμό, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο που είναι αυτό το οποίο έχει κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, την οικονομία που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο του εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο και φέρνει επομένω τεράστια ωφέλη στους πολίτες μας. <clears throat> Γι' αυτό χαιρετίζω ιδιαίτερα την άποψη που διατύπωσε ο πρώτος Λαμασούρ ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε και μια τέτοιου είδους ανάλυση θέμενες αξίες, για να γίνουν πιο σαφή τα ευρύτερα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μονάχα λοιπόν καθαροί και συνεισφορείς και αποδέκτες, αλλά τα ευρύτερα ωφέλη που παίρνουν οι χώρες μας από τη συμμετοχή σε μια ενιαία αγορά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κούλα, επίσης αναφέρθηκε και στο θέμα της τραπεζικής εποπτείας και στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ πρέπει να πω ότι εδώ έχουν γίνει κάποιες κοσμοϊστορικές αλλαγές. Το γεγονός ότι συμφωνήσαμε για μια ενιαία εποπτική αρχή και ενιαίο μηχανισμό εποπτείας η διάρκεια και η ένταση των διαπραγματεύσεων κατέδειξαν πόσο δύσκολο ήταν να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρειάστηκε να δώσει εντολές στους υπουργούς ΕΚΟΦΗΝ δύο φορές να συζητήσουν για μια συμφωνία επί των λεπτομεριών και όλα αυτά ήταν ιδιαίτερα κατεπήγοντα γιατί είδαμε πραγματικά τα όρια της εθνικής εποπτικής δραστηριότητας για τον τραπεζικό τομέα. Είδαμε ότι η χρηματοπιστωτικές αγορές είναι απόλυτα ολοκληρωμένες, αλλά η εποπτεία ασκείται μονάχα στα στενά εθνικά όρια. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό πια. Είναι πολλά τα διακυβευόμενα και ήταν σημαντική και ιστορική αυτή η απόφαση. Φυσικά θα εργαστούμε ως Κομισιόν για να προσθέσουμε τους δύο πρόσθετους πυλώνες που είναι απαραίτητοι στην ε, ενιαία εποπτεία. Καταρχήν τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Επίλυσης και επίσης τον Μηχανισμό Εγγύησης των Τραπεζικών Καταθέσεων. Από τη στιγμή που έχουμε κοινό νόμισμα, πιστεύουμε, από τη στιγμή που έχουμε κοινέ πολιτικές και έχουμε αυτή τη διαδικασία συντονισμού εξάντε, όλα αυτά θα είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουμε ότι το ευρώ θα γίνει το δεύτερο μεγαλύτερο διεθνές νόμισμα και θα είναι καλά ελεγχόμενο και με σωστή εποπτεία. Το θέμα της λογοδοσίας, της δημοκρατικής λογοδοσίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. <clears throat> Γι' αυτό η Κομισιόν έχει πει ότι είναι απαραίτητη η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως σε όλα τα θέματα που άπτονται της τραπεζικής εποπτείας. Επίσης, ένα από του λόγου που χρειαστήκαμε τόσο πολύ καιρό για να καταλήξουμε στη σωστή λύση για τον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό ήταν το γεγονός ότι οι Υπουργοί Οικονομικών είχαν εξετάσει με ιδιαίτερα λεπτόλογο τρόπο ποια ήταν η βέλτιστη κατανομή εξουσιών μεταξύ των εθνικών εποπτών και του ευρωπαϊκού επόπτη. Νομίζω ότι έχει βρεθεί η σωστή ισορροπία. Όλες οι χώρε έχουν δεχθεί αυτή τη λύση και τα εθνικά κοινοβούλια διατηρούν πολύ μεγάλη σημασία και δυνατότητες για τον έλεγχο των εθνικών υπο, εποπτικών αρχών. Είναι τόσο σημαντικός αυτός ο τωρέας που δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει κάποιο είδους αντιπαράθεση μεταξύ των εθνικών υποπτών και του, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όταν συζητάμε για θέματα ευρωπαϊκού επίπεδου. Έχουν ληφθεί δε όλες οι προφυλάξεις ώστε το σύστημα αυτό το οποίο εισήχθη είναι σωστά ζυγισμένο και εξασφαλίζει τι απαραίτητε ισορροπίε. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρω αυτό το σύστημα. Και αυτή είναι και μια απάντηση στον κύριο Χουάνγκ Γκόγκ, ο οποίο αναφέρθηκε και αυτό ω ένα από του τελευταίους ομιλητέ. Για τι άμεσε πληρωμές, όπω είπε ο συνάδελφο από την Λετωνία. Ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο θέμα, το οποίο εγείρεται κυρίως από τα νέα που πιστεύουν ότι η πρόοδος προς το τελικό στάδιο όταν οι άμεσες πληρωμές θα έχουν εξισωθεί μέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> θα μπορούσε να επιτευχθεί ταχύτερα. Βλέπουμε όμως και τώρα με τις διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές ότι ο ρυθμός προόδου περιορίζεται από τις δυνατότητες που έχουμε και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις, τους περιορισμούς σε επίπεδο προϋπολογισμών. Οι προτάσεις μας λοιπόν αντανακλούν αυτές τις διαφορές αλλά και τις προσπάθειες να κάνουμε το μέγιστο μέσα στις τωρινές δυνατότητες του προϋπολογισμού. Υπάρχει ένα ακόμα επιχείρημα το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να αναφερθεί. Είναι το γεγονός ότι τα νέα κάτι μέλη έχουν ευνοηθεί πολύ από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν δούμε λοιπόν τη συνολική υποστήριξη προς τους γεωργούς θα πρέπει να δούμε και το επίπεδο των άμεσων πληρωμών αλλά και το επίπεδο υποστήριξης για την αγροτική ανάπτυξη και τότε αν κάνουμε μια διαίρεση ανά εκτάρια τα πράγματα για τα, τα νέα κράτη-μέλη φαίνονται κάπως καλύτερα. Αλλά συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για να υπάρξει και η πληρέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Κύριε Τσούποφ, επίσης μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκών Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αν θέλετε θα το συνέδε αυτό και με το ερώτημα του κ. Σερβάς για την γενική διαφάνεια σε σχέση με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Ξέρω ότι αυτό είναι θέμα και στις Ολλανδία γιατί το ίδιο ερώτημα μου ετέθηκε εκεί. Όπω καταλαβαίνετε είναι δύσκολο για μένα να μιλήσω εξ του Συμβουλίου, αλλά εγώ εκπροσωπώ εδώ την Κομισιόν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων όπου προετοιμάζεται η κάθε διάσκεψη κορφή. και είναι γεγονό ότι ορισμένε φορέ για να μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία στο επίπεδο του Συμβουλίου θα πρέπει να βασιστούμε και στην πολιτική διέστηση του Προέδρου του Συμβουλίου υπό την αιγίδα του οποίου συντάσσονται τα συμπεράσματα των Συμβουλίων. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι εκπρόσωποι των ε, κρατών μελών στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συζητούν διαμακρών και με μεγάλη λεπτομέρεια τα θέματα αυτά παρουσία του κυρίου Φαν Ρομπάη και όλο και περισσότερο ένα τμήμα των συζητήσεών μας ε, γίνεται δημόσιο και παρουσιάζεται από τα κανάλια κτλ. Φυσικά και εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη αναμετάδοση από τα εθνικά κανάλια για τα θέματα αυτά. Σε σχέση με την ηλιοτυπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έχουμε τη φιλοδοξία ούτε την προσδοκία ότι η πρόταση της Κομισιόν θα γίνει δεκτή αμέσως και χωρίς αντιδράσεις. Υπάρχει πρόταση Κομισιόν εδώ και πολύ καιρό. Ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει προχωρήσει σε επίπεδα τα οποία δεν ήταν καν διανοητά πριν από μερικά χρόνια, μετά πριν από ένα ή δύο χρόνια. Αυτή η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν για το μέλλον ήταν ένα έγγραφο που είχε σαν στόχο να δώσει έναυσμα στη συζήτηση. Έχει γίνει αυτό και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η συζήτηση και θα θέλαμε να παρουσιάσουμε και σε εσά το φθινόπωρο αυτού του έτους ένα έγγραφο που αποτελεί το γενικότερο όραμα της Κομισιόν δεν είναι μονάχα τα οικονομικά και νομισματικά θέματα σε πιο μακρόπνο επίπεδο, αλλά το θέμα της μελλοντική ε, εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής ένωσης ως απόλυξη. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πιστεύω θα είναι μια μεγάλη ε, προβληματική, ένα σημαντικό θέμα για τις ευρωεκλογέ του 2014 και ελπίζουμε ότι το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η νέα Κομισιόν που θα διαμορφωθεί θα έχουν πράγματι μια σαφή εντολή από τους πολίτες για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε σε σχέση με αυτό το όραμα και το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια ολοκλήρωσης. Σε ό,τι αφορά τα θέματα διαφάνειας, προσπαθούμε να κάνουμε ότι μπορούμε περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, τις διάφορες ε, συναντήσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων, τα πρακτικά ή τις ε, μαγνητικές καταγραφές των αποφάσεων και των συζητήσεων. Μπορώ να σας δώσω ένα μακρό κατάλογο για αυτά τα οποία έχουν γίνει και μπορώ να σας δώσω αυτές τις πληροφορίες στα Εθνικά Κοινοβούλια, ποιες είναι οι βελτιώσεις που έχουμε επιφέρει για την μεγαλύτερη διαφάνεια του έργου της Κομισιόν και εμείς χαιρετίσουμε βέβαια και τις δικές σας προτάσεις για το τι θα μπορούσαμε να πράξουμε περισσότερο. Ο κύριος Νεκρό μίλησε για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Έχει δίκιο <clears throat> ότι αυτό είναι ένα απόσπαστο τμήμα όλων των συζητήσεων που κάνουμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εμεί μαθαίνουμε πολλά από τις συζητήσεις αυτές στην Κομισιόν. Αυτό το οποίο προσπαθούμε τώρα να επιτύχουμε είναι πρωτού προβούμε σε μια νομοθετική πρόταση να κάνουμε μια πλήρη εκτίμηση αντικτύπου με το πρίσμα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 30% των αποφάσεων της ε, ομάδας που κάνει τον έλεγχο αντικτύπου οδηγούν στο να ξαναγυρίσουμε <clears throat> στα Εθνικά Κοινοβούλια και να λάβουμε υπόψη τις απόψεις τους και σας διαβεβαιώ ότι θα στέλνουμε πάντα τις προτάσεις μας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και την έκθεση ε, αντικτύπου που περιλαμβάνει την εκτίμηση αναλογικότητας και επικουρικότητας και χαίρομαι που όλο και περισσότερες ε, απόψεις έρχονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια ως τμήματα του πολιτικού διαλόγου ή του ελέγχου της επικουρικότητας και δυστυχώς πολλές φορές καθυστερεί αυτή η διαδικασία πολύ περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε και δεν σας δίνουμε αμέσω άμεσες απαντήσει στα ερωτήματά σας. Τέλος, ο κύριος Λέιντεν, ο γερουσιαστής από την Ιρλανδία, έθεσε το θέμα της επικοινωνίας. Όλοι μας θα πρέπει να συνεργαστούμε για πιο θετική επικοινωνία. Δεν θέλουμε να παρουσιάσετε μονάχα η αρνητική εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάνουν πολλά μέσα ενημέρωσης, αλλά θα πρέπει να προβάλλουμε και τα θετικά στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει και πολλοί από εμά Εργαζόμαστε σκληρά τα τελευταία δύο-τρία χρόνια για να ξεπεράσουμε την κρίση. Ξέρουμε πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα αυτό για την Ιρλανδία και εμεί μπορώ να πω ότι έχουμε εντυπωσιαστεί τα μάλλα από τι προσπάθειε που κατέβαλαν οι Ιρλανδοί και η Ιρλανδική κυβέρνηση για τη σωστή εκτέλεση του προγράμματο <clears throat> σταθεροποίηση και με την ε, πρόπτικη να επανελθεί πολύ γρήγορα η Ιρλανδία στι αγορέ και πιστεύουμε ότι θα επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα με θετικό τρόπο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς. Ε, παρατήρησα ότι ε, λάβατε υπόψη την πρόταση για την τηλεοπτική μετάδοση των συζητήσεων της ε, Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν στενά για να κάνουν πραγματικότητα αυτή την εξαιρετική ιδέα. Πριν δώσω τώρα το λόγο στους Προέδρους των Αντίστοιχων Επιτροπών, θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου, Colin Barrett, για τις ε, τελειωτικές του ε, παρατηρήσεις. Ήθελα απλά να σχολιάσω σε σχέση με τα όσα είπε ο Βέλγος συνάδελφος για την ε, έλλειψη βάσει εθνικών κοινοβουλίων σε ευρωπαϊκά θέματα. Θέλω να το τονίσω και εγώ και μία από τις προτάσεις που εγώ έκανα ήταν να κάνουμε μια προσπάθεια να συμφωνήσουμε μεταξύ όλων των εθνικών κοινοβουλίων ότι σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία κάθε ίσως δύο μήνες όλα τα εθνικά κοινοβούλια θα συζητούν τα ευρωπαϊκά ζητήματα τα οποία εξετάζονται τη συγκεκριμένη στιγμή ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν αυτό γινόταν σε όλη την Ευρώπη και μπορούσε να υποστηριχθεί ε, ως Ευρωπαϊκή ημέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τώρα πώς αυτό θα υλοποιηθεί ίσως είναι πιο δύσκολο. Πιστεύω ότι ένα από τα προβλήματα συναντήσεων σαν αυτή είναι ότι ακούγονται πολλές καλές προτάσεις. Αλλά αναρωτιέται κανείς που καταλήγουν μετά το πέρας των συζητήσεων. Εγώ πιστεύω ότι Καλό θα ήταν να βρούμε έναν τρόπο προσαρμογής και υποστήριξη των καλών αποφάσεων εδώ και παρακολούθησής τους, ώστε να μην τις ξεχνάμε όταν εγκαταλείπουμε αυτή την αίθουσα. Εγώ θα ήθελα σοβαρά να ζητήσω από τα Εθνικά Κοινοβούλια να συζητούν τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ενδεχομένως μία μέρα το μήνα ή κάθε δίμηνο, να βρούμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε. Το μόνο που εγώ μπορώ να σκεφτώ είναι να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια τέτοια πρόταση σε συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ώστε όλοι οι αρχηγοί κυβερνήσεων και κρατών να συμφωνήσουν γι' αυτό. Πρέπει να ληφθεί η σχετική απόφαση, όχι απλά να το αφήσουμε να εωρείται και να ελπίζουμε ότι κάποια μέρα θα συμβεί. Πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία. Διότι εμεί, στα Εθνικά Κοινοβούλια, όσοι από εμά είμαστε μέλη μιας ε, Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, πράγματι δεν γνωρίζουμε καθόλου τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκά θέματα. Διότι αν οι εκθέσεις δεν ε, παρουσιάζονται στις Ολομέλειες, πώς να το γνωρίζουμε. Πραγματικά υπάρχει έλλειμμα εδώ και νομίζω ότι κάτι θετικό σε αυτό που προκύπτει από διασκέψαν αυτήν θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ένα σχόλιο για τον Γερμανό συνάδελφο που μίλησε για δημοψηφίσματα. Η Ιρλανδία, όπω ξέρετε, είναι ειδική στα δημοψηφίσματα, επειδή έχουμε ένα γραπτό σύνταγμα με πολλά λόγια. Και κάθε φορά που γίνεται αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εμεί πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα. είναι ιδιαίτερα μεγάλη ικανοποίηση όταν είναι επιτυχή. Αλλά είναι δυσάριστη η διαδικασία διότι όλοι όσοι αντιτίθενται στην έννοια της Ευρώπης ε, ξεκινούν σκηνοτενείς συζητήσεις ε, με πολλά θέματα που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το θέμα για το οποίο γίνεται το δημοψήφισμα. Ωστόσο αποτελεί τεράστια ανταμοιβή αυτή η επιβεβαίωση των λαών, του λαού που πολλές φορές έχουμε βιώσει. Η μόνη δυσκολία που εγώ διακρίνω όσον αφορά την τακτική διεξαγωγή δημοψηφισμάτων είναι ότι το, η προσέλευση είναι σχετικά χαμηλή το οποίο μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στην πολιτική πρέπει να το αναγνωρίσουμε ως μια δυσκολία επικοινωνίας δυσκολία κατανόησης της σπουδαιότητας των ζητημάτων Αυτά τα δύο ήθελα να σχολιάσω. Εγώ δεν φοβάμαι τα δημοψηφίσματα. Θεωρώ ότι πρόκειται μια εξαιρετική άσκηση, ειδικά όταν πετυχαίνει κανεί το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Επίση, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον Βέλγο συνάδελφο. Πρέπει να κάνουμε κάτι θετικό ώστε στις ολομέλειες όλων των εθνικών κοινοβουλίων να παρουσιάζονται σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα γιατί αν δεν συζητώνται εκεί πώς μπορούμε να απαιτούμε από το κοινό να τα καταλάβει. Τέλος, ε, κάτι άλλο που θεωρώ δύσκολο για το κοινό είναι η χρήση ορισμένων μορφών ευρωπαϊκής γλώσσας όπως το 2-pack και το 6-pack. Θεωρούμε δεδομένο ότι το κοινό γνωρίζει τι είναι το 6-pack και τι είναι το 2-pack και μερικές φορές ε, νομίζουμε ότι μιλάμε για ένα 6-pack ε, μπύρες, για ένα... μια εξάδα κουτάκια πρέπει να προσέχουμε όταν συζητάμε αυτά τα ζητήματα εκτός ενός φόρουμ σαν αυτό να μην θεωρούμε δεδομένο ότι ο κόσμος καταλαβαίνει με σαφήνεια γιατί συζητάμε. Ναι, ανακαλύψανε μάλιστα τα spread, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω, όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος Σούλτς, ότι σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο έχουμε την Europol TV που έχει στρατηγικές συνεργασίες με πολλά περιφερειακά, τοπικά, εθνικά, κοινοβουλευτικά, τηλεοπτικά κανάλια σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να φέρνει τους Ευρωπαίους πολίτες πιο κοντά στα όσα πράττουμε εδώ στην Ευρώπη και ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μας ευχαριστούσε ιδιαίτερα να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία και να δούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να εξοικειωθούν περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες με τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού, της ε, Επιτροπής Απασχόλησης, δεν ξέρω ποιος θέλει το λόγο, ο κύριος Λαμασούρ, Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Μερικά στοιχεία μόνο, έτσι, αποσπασματικά απαντήσεων ε, για, στις ερωτήσεις των εθνικών βουλευτών. Η Μπετίνα Κούντλα, της ΣΕΝΤΕΟΥ. Εδώ είστε. Έφυγε. Α, μάλιστα. Απλώς ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις, να συμπληρώσω τα λεγόμενα του Προέδρου Μπάρετ για ε, την προβληματική των δημοψηφισμάτων. Ρώτησε η Μπετίνα γιατί να φοβόμαστε τα δημοψηφίσματα. Μα είναι σαφές ότι αν ο, ο καγκελάριος Κόλ το 1992 είχε υποβάλει σε δημοψήφισμα τη συνθήκη του Μαστρίχτ και στρέφομαι προς τους Γερμανούς συναδέλφους, η πλειοψηφία θα ήταν αντίθετη με τη δημιουργία του ευρώ στη Γερμανία. Ο γερμανικός λαός, ωστόσο, είχε την ευκαιρία να αποφανθεί στις επόμενες εκλογές. Γενικέ και εκλογέ, ε, έβγαλε με τα τζάρουχια τον ε, καγκελάριο Κόλ. Κάθε χώρα μας έχει τις παραδόσεις της στη Γαλλία. Από τότε που αποχώρησε από την εξουσία ο, ο στρατηγός Ντεγκόλ, χάνοντας ένα δημοψήφισμα, το δημοψήφισμα θεωρείται ε, υπέρ ή κατά ε, ψήφισμα ε, εκείνου που κυβερνάει. Όταν είμαι εγώ στην εξουσία ε, παρακαθήμενη, καταψηφίζω οποιοδήποτε δημοψήφισμα και όταν εκείνη στην εξουσία καταψηφίζω εγώ. Προσοχή λοιπόν στη χρήση της άμεσης δημοκρατίας. Οι βουλευτές γνωρίζουν πολύ καλά ε, ποια είναι η ποιότητα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε σχέση με την άμεση δημοκρατία. Θα πρέπει να συνδυάζονται, αλλά κάθε χώρα έχει τις εθνικές της παραδόσεις. Απαντώντας ε, στο σχόλιο της κυρίας Κούντλα, το οποίο ακούμε συχνά, ε, που λέγει «Μα γιατί να αυξηθεί ο κοινοτικό προπολογισμό αφού έχουμε πλεόνασμα πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ, κονδύλια που δεν έχουν απορροφηθεί». Αυτό που ονομάζεται στη δική μας έτσι, γλώσσα που καταγγέλει ο πρόεδρος Μπάρετ στην Ευρωδιάλεκτο, ε, τα ε, υπόλοιπα προς εκαθάριση. Πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι ψευδό υπόλοιπα, ψευδό πλεονάσματα. Όταν ε, τίθενται σε ισχύ νέα προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα συνοχής, περιφερειακής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής, Χρειάζονται περίπου 18 μήνες σε κάθε κράτος μέλος για να στηθούν οι διαδικασίες, τα κριτήρια και τα έργα. Ε, ιδιαίτερα σε χώρες που είναι ομοσπονδιακού χαρακτήρα. Γι' αυτό αυτή η καθυστέρηση, αλλά είναι τεχνικής φύσεως των 200 δις. Δεν είναι ε, ε, αναπορόφητα κονδύλια πολιτικά, είναι τεχνικό το ζήτημα. Και ο επόμενος ομιλητής ε, από τη Λετωνία ανησύχησε από τις ανετικές επιπτώσεις που θα είχε αυτό για πούμε, τα κονδύλια συνοχής για τη χώρα του σύμφωνα με κάποιες περιόδους αναφοράς του παρελθόντος. Θα ήθελα ιδιαίτερα να χαιρετήσω την ε, παρέμβαση του κυρίου Σερβά, συναδέλφου από τις κάτω χώρες, που καταγγέλει και παραπονιέται για έλλειψη διαφάνειας. Και θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτόν τον καιρό προσπαθεί να σφετεριστεί την εξουσία. Ε, παραβιάζοντας ε, το πνεύμα των συνθήκων. Και πολύ ε, σημαντικά, δυστυχώς έχει αποχωρήσει ο πρόεδρος Βαρόν Πόη για να ακούσει τα λεγόμενά μας τώρα, αλλά ελπίζω να του διαβιβαστεί αυτό. Τι ορίζουν οι συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ως ρόλο να χαράσει τις μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές και τους προσανατολισμούς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Συμφωνούμε όλοι και χαιρόμαστε γι' αυτό γιατί όταν ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές της κρίσης χρέους, και ευτυχώς που υπήρχε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ευτυχώς που αντέδρασε και ευτυχώς που έσβησε την πυρκαγιά και επινόησε ευρηματικές λύσεις. Πολύ ωραία. Αντίθετα όμως, από εκεί και πέρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει την τάση να θεωρεί ότι είναι το ύψιστο όργανο και αυτή τη στιγμή έχουν συμφωνήσει τα μέλη του αυτό έχει ισχύ νόμου για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκείνη τη στιγμή ακριβώς, μάλιστα την επόμενη φορά, την άλλη εβδομάδα, αυτό τον καιρό έχουν στόχο να αποφασίσουν και να καθορίσουν τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές στον κοινοτικό προϋπολογισμό 2014-2020. Και αν συμφωνήσουν και ομόφωνα θα στραφούν σε εμά τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς εμάς με Y, τα Εθνικά Κοινοβούλια και να σας πούν ορίστε θαύμα Θαύμα! Συμφωνήσαμε, σώνεται η Ευρώπη για 10 χρόνια και βεβαίως πολιτικά συμφωνείτε, είστε υποχρεωμένοι να το δεχτείτε, να το κυρώσετε. Και στα Εθνικά Κοινοβούλια θα πούν ότι είναι ευρωπαϊκή απόφαση και σε εμά θα πούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι κοιτάξτε έγινε τέτοιο θαύμα, τώρα εσείς δεν μπορείτε να ανατρέψετε και να ε, παρεμποδίσετε αυτή την τεράστια πρόοδο για την Ευρώπη. Πλην όμως, επί της ουσίας εξακολουθούν να εργάζονται με όρους διαπραγμάτευσης διεθνούς ε, σύμβασης και συμφωνίας, όπως κάνουν οι διπλωμάτες, εγκρυπτό και παραβίστο, ενώ πρόκειται για τον προπολογισμό που είναι η πιο σημαντική πολιτική για τα κοινοβούλια που απαιτεί δημοκρατική συζήτηση πλήρως ειλικρινή, ανοιχτή, δημόσια, ο καθένας να εξηγεί και τα επιχείρηματά του και την ψήφο του και ε, η τελική ψήφος εναπόκειται στους ερετούς εκπροσώπους των λαών που γι' αυτό έχουν εκλογεί. Είναι σαν να έρχονται οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων στη Γερμανία για να αποφασίζουν για την επόμενη δεκαετία το γερμανικό προπολογισμό στο σύνολο τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Αυτό είναι σκάνδαλο και αμέσω το ανάτο δικαστήριο τη Καζρούη θα το εκείρωνε. Λοιπόν, ε, ε, βαίνουμε προ μία εκτροπή τη ε, κοινοτική λειτουργία και από πλευρά δημοκρατική είναι τελείω απαράδεκτη αυτή η εκτροπή απαράδεκτο τελείως και ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα συντονίσουμε τη δράση και την αντίδρασή μας στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό. Και εδώ συμφωνώ με την πάρα πολύ ωραία πρόταση του κυρίου Πρόεδρου Μπάρνετ να δούμε τι συνέχεια μπορούμε να δώσουμε στη σημερινή μας συνεδρίαση και να φροντίσουμε τις επόμενες συνεδριάσεις ε, να είμαστε ε, προετοιμασμένη με πολύ μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαμασούρη, κυρία Μπερές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για όσους παραμένουμε στο τέλος αυτής της ε, συνάντησης. Πραγματικά και εγώ συμφωνώ με την απογοήτευση του Βρετανού συναδέλφου. Την απογοήτευση που εξέφρασε για την απουσία του κ. Βανδρομπέη, του κ. Μπαρόσο, παρότι χαίρομαι για την ε, παρουσία του κ. Σεύκοβετς και τη κυρίας Ποδηματά. Σε αυτό το debriefing, όπω μα έχουν μάθει να κάνουμε Βρετανοί, θα πρέπει να σημειωθεί αυτό το σημείο. Αυτό που ξεκινήσαμε φέτο θεματικές πρώτα απ' όλα συνεδριάσεις ε, παράλληλες επέτρεψαν σε περισσότερους συναδέλφους να εκφραστούν χωρίς ε, να έχουν προετοιμάσει έγγραφα. Μας επέτρεψαν μεγαλύτερη αλληλεπίδρες και πιο βαθιές συζητήσεις σε αυτά τα εργαστήρια. Πιστεύω επίσης ότι αυτή η ιδέα του να έχουμε τους προέδρους των τριών ε, θεσμικών οργάνων στο τέλος της άσκησης είναι πολύ καλό γιατί αυτό επιτρέπει να φέρουμε την εργασία σε ένα απαραίτητο επίπεδο και να περάσουμε το μήνυμα, αλλά η εκ των ονουκάνευ συνθήκη είναι να παραμένουν οι πρόεδροι αυτών των τριών θεσμικών οργάνων μέχρι το τέλο τη ανταλλαγή απόψεων. Μάλιστα, ακόμη περισσότερο επιδιορισμένα μηνύματα που εμεί προσπαθούμε να περάσουμε είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να τα ακούσουν. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο Μπάρετ. Πιστεύω ότι και οι δύο του ομιλίε. Ε, ήταν εξαιρετικά σαφής, εξαιρετικά θετική η συμβολή του για τη συνέχιση των εργασιών μας και για να κατανοήσουμε βάσει και των όσων είπε ο πρόεδρος Μαρτίν Σουλς χθες στο δείπνο το πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ο καθένας μας πρέπει να έχει στο νου του το δημοκρατικό ορίζοντα αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε να κάνουμε δουλειά στις χώρες μας. Οι προτάσει που κάνατε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις κοινοβουλευτικέ εργασίες μου φαίνονται και με βέβαιοι ε, πολλά υποσχόμενε για το μέλλον. Θα ήθελα να επανέλθω αυτή την τελική ομιλία στην ιδιαίτερη φύση τη άσκηση αυτή εδώ που ουσιαστικά αποτελεί την κατάληξη μιας διαδικασία που έχει ξεκινήσει πριν πολύ καιρό και την αφετηρία μιας άλλης διαδικασία. αυτό το ευρωπαϊκό εξάμενο και η ετήσια ανασκόπηση της ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να θυμόμαστε τι μας λένε οι συνθήκες όσον αφορά τον ανταγων... την αρμοδιότητα όσον αφορά την οικονομική και νομισματική πολιτική και τι ορίζουν οι συνθήκες για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Αυτοί είναι τομεί που δεν μπορούμε να θεωρούμε ένα copy-paste των όσων κάναμε στην εξωτερική πολιτική. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες των μεν και των δε είναι πολύ διαφορετικές. Δεν μπορούμε να παραλληλήσουμε τους ε, αντίστοιχους μηχανισμούς. Η δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω για το τι μπορούμε να κάνουμε μαζί με τον Αλάν Λαμασούρ και νομίζω ότι σε αυτή την αίθουσα είμαστε από τους λίγους που είχαμε αυτό το διπλό προνόμιο να συμμετέχουμε στις ε, συνθήκες. Ε, στη συνθήκη υπήρχε δυνατότητα συγγραφής του κειμένου μαζί. Είχε τεθεί το ζήτημα της νομιμότητας. Μιλούσαμε για μια διακυβέρνηση πολλών επιπέδων σε πραγματικό χρόνο. Στην άσκηση της αιτήσιας επισκόπησης της αναπτύξης και του Ευρωπαϊκού Εξαμένου θεωρώ ότι δεν μπορούμε όλοι μαζί να γράψουμε ένα ψήφισμα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το έρινο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ίσως κάνω λάθος, αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να ζυγίσουμε όλες αυτές τις ε, απόψεις για να τις ε, στείλουμε στο έρινο Συμβούλιο. Θα πρέπει να δούμε πώς... Ε, είναι εξαιρετικά πολύτιμες οι ανταλλαγές που κάναμε σε αυτήν εδώ την εκδήλωση και υπό αυτό το πνεύμα όπως ανέφερε ο κύριος Μπάρετ πρέπει να δούμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε στο μέλλον. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω, διότι πιστεύω η ουσία υπόθηκε σε αυτές τις τρεις τελευταίες μέρες που περάσαμε μαζί και χαίρομαι ιδιαίτερα που με όλο τον πλούτο που αποκομίσαμε φέτος θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να επαναλάβουμε την διακδηλώση του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευχαριστώ ο κύριος Σεύκοβιτς για τις τελευταίες του παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ νιώθω ότι με ενθαρρύνει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση που έχει λάβει η χώρα <clears throat> με, από τη Δευτέρα παρακολουθώ αυτήν την συνδιάσκεψη και ήταν σαφής και η θέση της Ιρλανδίας ότι πρέπει να ενισχυθεί η διακοινοβουλευτική συζήτηση και ο συντονισμός γιατί είμαστε τώρα στη φάση της περαιτέρω εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα εξασφαλίσουμε την κατάλληλη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο δίδαγμα το οποίο αντλώ από αυτές τις τρεις μέρες είναι ότι πρέπει να προβούμε σε καλύτερο συντονισμό, ιδίω στον τομέα τον κοινωνικό και να επιτύχουμε και μεγαλύτερη σύγκληση στα θέματα αυτά. Πάρα πολύ είναι σημαντικό αυτό, γιατί αλλιώς <clears throat> κινδυνεύουμε να έχουμε όλο και πιο έντονο ανταγωνισμό προς τα κάτω και θα θέσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό υπόδειγμα σε κίνδυνο. <clears throat> Νομίζω ότι η πρόταση της Μπερές που εγώ αναφέρω σε κάθε Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων το να μπορούν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια γενναία νέων Ευρωπαίων που πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και στη δημοκρατία και στην ικανότητά μας να παίρνουμε σωστές αποφάσεις, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε χωρίς καμιά ελπίδα κατάρτισης ή θέσης απασχόλησης. Ένα ακόμα στοιχείο για τα μη δαπανόμενα, τα μη εκταμιευόμενα ποσά. Υπάρχουν σε πολλα κατημέλη τέτοια ποσά λόγω διαδικασιών που δεν είναι πάντα με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά χρειάζεται να έχουμε και λογικούς ετήσιους προϋπολογισμούς. Είναι δύσκολο να δαπανίσει κανείς ένα κονδύλιο αν οι προϋπολογισμοί υποπροϋπολογίζουν τα ποσά τα οποία χρειάζονται. Μεταφέρονται τελικά <clears throat> τα χρήματα με τον τρόπο αυτό στο τέλος της περίοδου δημοσιονομικών προοπτικών και είναι πολύ δύσκολο να δαπανηθούν από τα κάτι μέλη είναι απαραίτητο να υπάρχει ποιότητα εκταμείευση και επίση σωστή προπολογισμοί σε αιτήσιο επίπεδο που σέβονται τι δημοσιονομικέ προοπτικέ, αλλά να είναι ρεαλιστική η προπολογισμοί αυτή. Και το τελευταίο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να σα αναφέρω είναι το εξή. Πιστεύω ότι οι δύο αυτές αρχές που πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον είναι πολύ σημαντικέ. Πρώτα απ' όλα το να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει λογοδοσία στις αποφάσεις, για τις αποφάσεις στο επίπεδο όπου λαμβάνονται, αλλά και εκεί που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο αυτές οι αποφάσεις και συγχρόνως να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση ανάλογη με το βαθμό εκχώρησης εξουσιών από τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με καλή θέληση και με την ευελιξία και δημιουργικότητα που φάνηκε στο Δουβλίνο και στις Βρυξέλλες τελευταίες μέρες, θα μπορέσουμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε την Πρόεδρε, κύριε Σεύκοβιτς. Αγαπητοί συνάδελφοι, στα αγγλικά και στα γαλλικά, νομίζω ότι έχουμε όλη επίγνωση ότι οι συζητήσεις που διοργανώνουμε στα πλαίσια της πρώτης ε, Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας για το συντονισμό και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο λαμβάνουν χώρα σε μια πάρα πολύ σημαντική συγκυρία ε, μετά τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας ε, επισκόπησης για την ανάπτυξη. Και όπως πολύ συχνά ακούστηκε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων μας κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αλλάζουν οι ε, αρμοδιότητες ε, με ε, νέες μεταρρυθμίσεις και θα αλλάξουν ακόμα περισσότερο για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων, για την οικονομική διακυβέρνηση. Πολλά κράτη-μέλη βλέπουν το ευρωπαϊκό επίπεδο να επεμβαίνει σε όλες τις πολιτικές σχεδόν, σε χώρες που εφαρμόζουν μνημόνια και ε, δυστυχώς αυτές οι χώρες βλέπουν να τους επιβάλλονται πολιτικές. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει βεβαίως. Για να δούμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα ε, των προγραμμάτων αυτών όταν επιβάλλονται έτσι στην εφαρμογή τους. Ε, ταυτόχρονα τώρα είναι κοινή πεποίθηση ότι το δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο προϋπήρχε έτσι και αλλιώς ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχει ε, επιδεινωθεί έτη περαιτέρω, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και συνεπώς είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να ε, φαίνεται και να ταυτοποιείται αυτός που λαμβάνει την απόφαση και φέρει και την ευθύνη τελικά για την υλοποίησή της. Οι συζητήσεις λοιπόν που είχαμε κατά τη διάρκεια του τριημέρου απέδειξαν ότι σε εμά εναπόκειται, εμά του ερετού εκπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είμαστε εθνικοί βουλευτέ είτε ευρωβουλευτέ. Είτε είμαστε στο Ευρωπαϊκό είτε στα Εθνικά Κοινοβούλια. Σε εμά λοιπόν εναπόκειται να βρούμε τους σωστούς, κατάλληλους τρόπους να συνοδεύουμε και να πλαισιώνουμε τις αποφάσεις ε, για την πολιτική ε, που δεν σέβονται πλέον ε, εθνικά σύνορα και θα πρέπει η κοινοβουλευτική διάσταση να ακολουθεί. Πολλά θέματα απομένουν να λυθούν ε, στα πλαίσια αυτού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και επίσης στα πλαίσια της εντολής του Δημοσιονομικού Συμφώνου ε, το περίφημο άρθρο 13, το οποίο γέννησε πολλές συζητήσεις, όπως γνωρίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, ε, πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια αυτού του τροιμέρου συζητήσεων κυριάρχησε ε, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, η κοινοτική προσέγγιση και χάρη στην ποιότητα των δικών σας παρεμβάσεων και των συζητήσεών μας και χάρη στην έκθεση και στις αναφορές που θα κάνουμε μάλλον ε, στους εκλογείς μας, πιστεύω ότι καταφέραμε να βελτιώσουμε κάπως ε, τη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Βεβαίως παραμένει ακόμα μακρύς ο δρόμος, αλλά είμαστε εμείς σε θέση να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας και την ποιότητα των παρουσιάσεων σας. Καλό σας απόγευμα.